Um, Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να ξεκινήσουμε τη συνεδρίασή μας γιατί ήδη έχουμε μια καθυστέρηση. I Σας παρακαλώ λοιπόν να καθίσετε. Σας ευχαριστώ πολύ. Να ξεκινήσουμε με το σημείο 1 της ημερήσιας διάταξης ε, να σας ανακοινώσω δηλαδή ότι όσοι ήθεστε ότι η συνεδρίασή μας είναι στο διαδίκτυο να σε ταυτόχρονη αναμετάδοση και επίσης θα θέλαμε να δούμε το θέμα της ε, κυρίας Μάνερ που θέλει αντί να παρουσιαστεί το θέμα της ε, στις 5 να το παρουσιάσει στις 3. Και όλες οι υπόλοιπες εκθέσεις λοιπόν θα ακολουθήσουν με κάποια καθυστέρηση. Επίσης να θυμίσω σε όλους ότι έχουμε μια πολύ γεμάτη μερίσια διάταξη και το κάθε σημείο το έχουμε ανακοινώσει σε κάποια συγκεκριμένη ώρα, αλλά μπορεί να υπάρξουν ε, απρόβλεπτες ε, καταστάσεις ε, και άρα κάποια σημεία να προφω... τα εξετάσουμε νωρίτερα ή αργότερα. Γιατί είναι σημαντικό, αν δεν είστε στην αίθουσα οι ίδιοι, κάποιος να παρακολουθεί τι γίνεται και αν πρέπει να μιλήσετε να είστε εγκαίρος στην αίθουσα, ώστε να μην χρειάζεται να καθυστερήσουμε για τις εισηγήσεις. Αυτά όσον αφορά την ημερήσια διάταξη και την έγκρισή τη. Δεν νομίζω να υπάρχουν αντιρρήσει, οπότε την εγκρίνουμε και περνάμε στο σημείο 2, που είναι η έγκριση των πρακτικών τη συνεδρίαση τη 26η Απριλίου και τη 8η ε, Μαου. Τα πρακτικά είναι διαθέσιμα, έχουν διανεμηθεί και θα θεωρήσουμε πώς εγκρίνονται στο τέλος της συνεδρίασης αν δεν έχετε υποβάλει εσείς ε, αντιρρήσεις. Ανακοινώσει του Πρόεδρου. Έχω δύο αρκετά σημαντικά πράγματα να σας ανακοινώσω. Το ένα είναι μικρό αλλά πολύ σημαντικό και θα ήθελα και η βοηθή να ενημερώσουν τους ευρωβουλευτές που δεν είναι παρόντες ότι η εκτύπωση των κειμένων καταρχήν κοστίζει και δεύτερον παίρνει πάρα πολύ χρόνο για τις υπηρεσίες. Οπότε μας ζήτησαν οι υπηρεσίες μας να κρατήσουμε για την επόμενη συνεδρίαση τα έγγραφα που διανεμήθηκαν σήμερα και κυρίως τους γενικούς κανονισμούς. Οπότε σας παρακαλώ να τα πάρετε μαζί σας, αλλά όχι σπίτι σας, στο γραφείο σας και να τα ξαναφέρετε όλα αυτά τα έγγραφα στις 11. Ο κύριος Βανίστελ Όσοι δεν τα διαβάζουν επίσης να τα φέρουν πίσω και να τα επιστρέψουν τα έγγραφα. Κοιτάξτε, δεν μπορώ να σας υποχρεώσω να τα διαβάσετε, αλλά τουλάχιστον να το πάρετε και να το φέρετε και πίσω ξανά. Και τώρα να περάσουμε στο επόμενο σημείο που αφορά την δημοσιονομική διαδικασία για τον προϋπολογισμό του 2013. Δυστυχώς δεν είμαστε η μόνη επιτροπή σε αυτή την κατάσταση. Υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά τις προθεσμίες για τις ε, τροπολογίες ε, περί προϋπολογισμού και την ψηφοφορία που έχει οριστεί στις 6 Σεπτεμβρίου. Ε, δεν θα έχουμε τον συνηθισμένο χρόνο για να περάσουμε από την φυσιολογική διαδικασία με την παρουσίαση εδώ, υποβολή τροπολογιών και γι' αυτό θα ήθελα να προτείνω το εξή. Την ίδια διαδικασία που χρησιμοποιήσαμε δηλαδή πέρυσι που σημαίνει ότι θα πρέπει να δείξουμε εμπιστοσύνη στους εισηγητές και στους στον ε, πρόεδρο της Επιτροπής Έχουμε έρθει σε επαφή με τον εισηγητή, τους σκιώδεις, τους συντονιστές και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να ακολουθήσουμε αυτή τη διαδικασία που θα είναι περίπου, όπως είπα και πέρυσι, θα αποτελείται από τα εξή. Πρώτα απ' όλα, η εντολή ε, εξοδοτεί τον Πρόεδρο και τον εισηγητή να τροποποιήσουν οποιασδήποτε περικοπές στην πρόταση της Κομισιόν που θεωρούν επαρκή και ότι ανταποκρίνονται επαρκής και ότι ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις. και να εξουσιοδοτήσουν τον Πρόεδρο και τον εισηγητή ότι αν το Συμβούλιο υποβάλει περικοπές Να έχουν την εντολή λοιπόν να επαναφέρουν το σχέδιο προπολογισμού της Κομισιόν. Δηλαδή να μην δεχτούμε τις πορικοπές σε αυτό το στάδιο. Ελπίζουμε να μην προτείνουν περικοπές, αλλά σε περίπτωση που προτείνει περικοπές το Συμβούλιο να μπορούμε να τις αρνηθούμε. Επίσης θα ήθελα να σας ρωτήσω, να σας ζητήσω να μας δώσετε εντολή ώστε να καταθέσουμε οποιοδήποτε πιλωτικό πρόγραμμα, προπαρασκευαστική δράση ή πρόγραμμα τεχνικής βοήθειας που συμφωνηθεί από τις πολιτικές ομάδες. Πάλι για τον εισηγητή και τον Πρόεδρο. Καθώς και την εντολή για να υποβάλουμε τροπολογίε στη θέση του Συμβουλίου, πράγμα που θα ήταν απαραίτητο για να προστατευτούν οι στόχοι τη πολιτική συνοχή σύμφωνα με τι διαδικασίε για το πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο και τι σχετικέ διατάξει τη διοργανική συμφωνία. Και φυσικά αυτέ οι τροπολογίε αν τελικά προκύψουν, θα τη συζητήσουμε με τους ε, συντονιστές και τους εισηγητές του προϋπολογισμού για το 2013. Και τελευταία παρατήρηση που θα ήθελα να δεχτείτε, πρόταση μάλλον, μετά από αυτή τη διαδικασία που σας παρουσίασα, ένα σχέδιο γνωμοδότησης για το ψήφισμα για τον προϋπολογισμό να υποβληθεί στην ε, συνεδρίαση του Ιουλίου και το αποτέλεσμα να ψηφιστεί στο Σεπτέμβριο, στις 13 δηλαδή μετά από την ψηφοφορία της Ολομέλειας. Γι' αυτό είναι η ειδική διαδικασία. Αν συμφωνείτε με όλα αυτά, μπορούμε να κλείσουμε αυτό το σημείο της ημερησίας διάταξης και να περάσουμε στο τρίτο σημείο, που είναι Γενικός Κανονισμός Κοινές Διατάξεις για τα Ευρωπαϊκά Ταμεία. Να σας ενημερώσω ότι έχει μεταφραστεί Επίσης έχουμε εργαστεί η γραμματεία, οι συγητές και οι βοηθοί τους έχουν εργαστεί για τον κατάλογο ψηφοφορίας. Δεν έχει ακόμα τελειώσει η δουλειά, αλλά κοντεύει, οπότε θα τελειώσουμε γέρος. Και θα ήθελα επίσης να πω ότι γίνεται η συζήτηση για το γενικό κανονισμό αυτή τη φορά χωριστά σε δύο μέρες. Δηλαδή, μία ώρα και ένα τέταρτο τώρα και θα έχουμε και άλλη μία ώρα αύριο για το ίδιο θέμα. Και η τρίτη πληροφορία είναι ότι για αυτή τη συζήτηση έχουμε καλέσει τον κύριο Μάρικ Βόσνικ που είναι ε, ε, εισηγητής της Επιτροπής των Περιφερειών για το κοινό στρατηγικό πλαίσιο ώστε να συζητήσει μαζί μας τη θέση της Επιτροπής των Περιφερειών και αν δεν σας ε, πειράζει θα ήθελα να ξεκινήσω με εκείνον για τη συζήτηση αυτού του σημείου. Οπότε κύριε Βόσνικ έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε κυρίες και κύριοι ευρωβουλευτές. Καταρχήν, σας ευχαριστώ για αυτή την πρόσκληση να μιλήσω σε αυτή την ε, συνεδρίαση της Επιτροπής Περιφερειακών ε, υποθέσεων αυτή τη στιγμή που συζητάμε το έγγραφο που υπέβαλε η Κομισιόν. Η Επιτροπή των Περιφερειών παρακολουθεί τις συζητήσεις με μέγα ενδιαφέρον και περίμενε την έκδοση αυτού του εγγράφου με μεγάλες προσδοκίες. Ελπίζουμε πως αυτό το πρόγραμμα θα είναι θετικό και για τις περιφερειακές κυβερνήσεις ή την τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί πρέπει να προτείνουν λειτουργικά προγράμματα. Από τη μια πλευρά λοιπόν το περιμέναμε αυτό το έγγραφο, από την άλλη όμως υπάρχει μια ανέστηση απογοήτευσης Θα θέλαμε λοιπόν να υιοθετήσουμε την τελική μας γνώμη για αυτό το θέμα τον Οκτώβριο. Υπό την ιδιότητά μου ως εισηγητής, θα πρέπει να τονίσω πως ε, η Επιτροπή των Περιφερειών έχει ήδη εγκρίνει έκθεση για το, χρηματοδότηση για τον γενικό κανονισμό και το κοινό στρατηγικό πλαίσιο θα είναι αντικείμενο μιας άλλης γνωμοδότησης. Επί τη βάση λοιπόν ε, ενδελεχούς και πλήρους διαβούλευσης με διάφορους ε, ε, δικαιούχους γιατί διοργανώνουμε διάφορες εκδηλώσεις και καθώς και φιλοξενήσαμε κάποιους από τους εταίρους μας στην Επιτροπή των Περιφερειών εδώ στις Βρυξέλλες. Είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε συζητήσεις με πολλούς εισηγητές τόσο στην Επιτροπή των Περιφερειών όσο και εδώ στο Κοινοβούλιο με την κυρία Πρέλ και τον κύριο Βανίστερ Ρόι. Έχουμε λοιπόν μια κάποια ιδέα αν δείτε την γενική εικόνα του τι προβλέπεται από την πρόταση της Κομισιόν, ο στόχος αυτής της πολιτικής συζήτησης φαίνεται να είναι ε, αυτό το γενικό στρατηγικό πλαίσιο να είναι χρήσιμο για την τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση ώστε να μπορέσουν να προτείνουν ε, προγράμματα εταιρική σχέσης. Εμείς καλωσορίζουμε το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τώρα αποτελεί ένα βασικό σημείο, για αυτές, ένα βήμα για αυτές τις διαπραγματεύσεις και ε, είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που η Επιτροπή των Περιφερειακών Υποθέσεων είναι η Περιφερειακής Ανάπτυξης είναι η Επιτροπή με την οποία συνεργαζόμαστε. Ε, διαβάσαμε το σχέδιο που συνέταξε η κυρία Κρέλου και ο κύριος Βανίστεροι και καταλάβαμε ότι, βλέπω ότι έχουμε κοινέ απόψεις για πολλά θέματα και ότι το έγγραφο αυτό περνά το περιεχόμενο της Επιτροπής των Περιφερειών. Η Επιτροπή των ε, Περιφερειών στηρίζει πλήρως την θέση του Ευρωκοινοβουλίου γιατί πιστεύουμε πως ε, ορισμένα σημεία θα πρέπει να αποτελούν παράρτημα και όχι πράξη κατά εξουσιοδότηση. Και εδώ συμφωνούμε. Τώρα όσον αφορά την ίδια την φύση του στρατηγικού πλαισίου θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την ιδιαιτερότητα της ε, τοπικής αυτοδιοίκησης σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολύ σημαντικό στοιχείο αυτό όσον αφορά την περιφερειακή αυτή προσέγγιση και τη δυνατότητα ε, σχηματισμού αυτών ε, των παρεμβάσεων ε, σε διάφορες περιοχές της Ευρώπης. Από την άλλη πλευρά θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή στους διάφορους μηχανισμούς συντονισμού. Αν λοιπόν αυτά τα πέντε κονδύλια και όλα τα άλλα μέσα ε, πρέπει να συμβιώσουν γιατί αυτή είναι η βασική προϋπόθεση εδώ, ο μηχανισμός συντονισμού θα πρέπει να είναι ξεκάθαρος. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει θέμα με τις ε, δράσεις κλειδιά και αυτές θα πρέπει να είναι ευρείες, ε, να έχουν ένα ευρύ χαρακτήρα. Και αν δείτε το έγγραφο της Κομισιόν, ε, όντως αυτό ισχύει. Πιστεύουμε λοιπόν ότι <clears throat> θα πρέπει να εξετάσουμε αυτά τα θέματα όσο γίνεται με πιο συνεπή τρόπο. Ο κατάλογος που μας παρουσιάζεται θα πρέπει να αποτελεί έναν ανοιχτό ε, κατάλογο. Γιατί αν ε, θεωρηθεί ως κλειστός κατάλογος ορισμένες ε, πρωτοβουλίες και προτάσεις που προκύπτουν προέρχονται από τις περιφέρειες θα μπορούσαν να παρεμποδιστούν. Συμφωνούμε με την ιδέα ότι τα κονδύλια ε, από το στατικικό πλαίσιο θα πρέπει να στηρίξουν την εφαρμογή των, της στρατηγικής Ευρώπη 2020, αλλά θα πρέπει να ξεπεράσουμε και αυτό το σημείο γιατί η συνθήκη σαφώς λέει ότι η οικονομική και η εδαφική συνοχή θα πρέπει να είναι ένας άλλος κύριος στόχος που θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας πάντα. Επιπλέον, θα πρέπει να εξετάσουμε την πολυθεματική προσέγγιση και δυστυχώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει ε, πετύχει πολλά πράγματα σε αυτό το τομέα και αυτό πρέπει να το τονίσουμε. Καλωσορίζουμε το γεγονός ότι στο έγγραφο τονίζεται και αναφέραμε εδώ στο έγγραφο που έχει συντάξει οι, που έχουν συντάξει οι της Επιτροπής ε, περιφερειακής ανάπτυξης ε, υπάρχουν διάφορα θέματα όπως και παράδειγμα το LIFE που είναι μια πολύ φρόσδεκτη ε, εξέλιξη ότι δηλαδή αυτά τα, το κονδύλια ε, όντως αναφέρονται εδώ. Επιπλέον θα ήθελα σύντομα να αναφέρω το θέμα της συγκεκριμένης επιχείρησης ή της... Ε, και των ολοκληρωμένων εδεφικών επενδύσεων που λείπουν από το κείμενο, ενώ στο παράρτημα υπάρχουν δύο. Η ανάπτυξη των τοπικών ε, κοινοτήτων αναφέρεται μόνο δύο φορές. Στηρίζουμε λοιπόν τα οριζόντια μέτρα για την καταπολέμηση των διακρίσεων και για την προώθηση της ισότητας των φύλων αλλά η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση φαίνεται να μην περιλαμβάνεται σε αυτό το έγγραφο και αυτό από την άποψη της Επιτροπής των Περιφερειών είναι πολύ σημαντικό. Διότι αυτή η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση είναι κάτι που θα χρησιμεύσει στο μέλλον. Επίσης, Καλωσορίζουμε την έμφαση που δίνεται στις δημογραφικές αλλαγές και στην πολυεπίπεδη διακυβέρνηση. Ε, στο κείμενο που χθε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τέλος κάποιες άλλες παρατηρήσεις που έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μάλλον που αφορούν το κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η Επιτροπή δεν αναφέρεται σε θέματα όπως οι πιο απομακρυσμένες από περιοχές, οι ορεινές περιοχές και άλλα. Τα σημεία αυτά λείπουν. Και ωστόσο πρέπει να γνωρίζουμε το γεγονός ότι αυτά τα σημεία είναι πολύ δύσκολα και πρέπει σαφώς να αναφέρονται με λεπτομέρειες. Τώρα, όσον αφορά τις προτεραιότητες συνεργασίας, αυτό που λείπει είναι οι μηχανισμοί για διεθνική συνεργασία. Και από την άλλη πλευρά, ε, συνεργασία με το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Είναι παράξενο αυτό. Μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο αυτή η διεθνική και περιφερειακή συνεργασία είναι κάτι που θα πρέπει διερκώς να έχουμε υπόψη, γιατί αυτού του είδους η συνεργασία είναι πολύ σημαντική. Τα σημεία αυτά λοιπόν θα πρέπει να επανεισαχθούν ή να εισαχθούν στο κείμενο της Κομισιόν. Όπως ίσως γνωρίζετε, η διαβούλευση μέχρι τώρα έχει οδηγήσει σε μια κάπως επικριτική στάση απέναντι στο έγγραφο της Κομισιόν που έρχεται σε αντίθεση με τη θετική μας ε, στάση απέναντι στο έγγραφο της Επιτροπής ε, ε, Περιφερειακής Ανάπτυξης και αυτό το σημείο θα ήθελα να το τονίσω γιατί αυτά όλα θα είναι αντικείμενο και κομμάτι της νομοδότησής μου προς την Επιτροπή των Περιφερειών. Ελπίζω λοιπόν πως με αυτόν τον τρόπο θα στηρίξουμε και τις συζητήσεις εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο και θα δείξουμε σαφώς ότι συμφωνούμε μαζί σας. Σας ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο. Μάλιστα, από συνάδελφοι θα πρότεινα να ανοίξουμε τη συζήτηση για το γενικό κανονισμό συμπεριλαμβανομένων των παρεμβάσεων που προέρχονται από την Επιτροπή των Περιφερειών. Οποιοδήποτε λοιπόν θέλει να μιλήσει, μπορεί να μιλήσει τόσο για τις τροπολογίες που έχουν κατατεθεί στο Κοινοβούλιο, όσο και για όσα μας είπε ο κύριος Βόσνιακ αρχίσουμε με τους εισηγητές για τον γενικό κανονισμό. Η Κωνσταντζα ήταν πιο γρήγορη από τον Λάμπερτ σήμερα. Σήκωσε πρώτη το χέρι της. Κωνσταντζα, λοιπόν, πρώτα εσύ. Ευχαριστώ, Ντανούτα. Ε, νομίζω, καταρχάς, και από μένα και από τον Λάμπερτ ε, αξίζει να ευχαριστώ σε όλους τους συναδέλφους ε, που με τόση μεγάλη ενέργεια εργάστηκαν και συνεργάστηκαν και θα συνεργαστούν στην ανάλυση του ε, συνολικού κανονισμού αλλά και στις, στα αποτελέσματα που οδήγησαν σε πάνω από 2.000 ε, τροπολογίες. Υπάρχει ένα ογκόλυφος πάνω στο τραπέζι μας. Νομίζω ότι δείχνει αυτό πόσο εντατικά δουλέψαμε τις τελευταίες εβδομάδες μετά από την πρώτη γρήγορη ματιά στις τροπολογίες μπορούμε να δούμε ότι πολλές ε, τροπολογίες πηγαίνουν προς μια παρόμοια κατεύθυνση. Ο ε, των περιφερειακών και τοπικών ε, αρχών, η ευελιξία, το αποθεματικό επιδόσεων, ε, θεματική συγκέντρωση, τα δικαιώματα των ε, ανθρώπων με δικές ανάγκες, όλα αυτά μπορεί να έχουν επιρροή στα διευθυντικά ταμεία, μηχανισμοί ελέγχου και απλούστευσης, όλα αυτά είναι σημεία τα οποία ε, συζητήθηκαν εντατικά και οι τροπολογίες νομίζω αντικατοπτρίζουν ακριβώς αυτή την κατεύθυνση για να είμαστε σίγουροι ότι έχουμε μια ισχυρή θέση στην ε, ψηφοφορία της 11ης Ιουλίου για το Κοινοβούλιο και με αυτόν τον τρόπο να έχει κανείς μια καλή εντολή διαπραγμάτευσης με την Κομισιόν. Νομίζω ότι στην ουσία οι τροπολογίες είναι επίσης το αποτέλεσμα μιας εντατικής εργασίας ε, το τελευταίο διάστημα. Συνεχώς ε, συζητούσαμε μεταξύ μας ε, πώς θα πρέπει να είναι η κατεύθυνση που θα ακολουθήσουμε για τη μελλοντική πολιτική συνοχής και πραγματικά ήταν πολύ κουραστικό για τους συμμετέχοντες αλλά ελπίζω ότι θα μας ανταμείψει το αποτέλεσμα και θα μπορέσουμε να δώσουμε ένα καλό σήμα με την ψηφοφορία τον Ιούλιο. Νομίζω επίσης ότι τον Ιούλιο όταν θα ψηφίσουμε θα στείλουμε και ένα πολιτικό σήμα ιδιαίτερα έντονο, ε, σημαντικό προς τα έξω. Θα είμαστε δηλαδή η πρώτη επιτροπή που ασχολήθηκε με αυτό το μεγάλο ε, πακέτο κανονισμών ε, για το 2014 με όλα, που έχει να κάνει με όλα τα προγράμματα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ένα μήνυμα που λέει ότι είμαστε έτοιμοι να δουλέψουμε, είμαστε ενεργοί και δεσμευόμαστε για τις περιφέρειες της Ευρώπης και δεν θέλουμε να διώξουμε από άνω μας τις δύσκολες διαπραγματεύσεις και αυτό γίνεται σε μια εποχή οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης ε, που με την πολιτική συνοχής θα μπορέσουμε να δώσουμε ένα εργαλείο επενδύσεων και ανάπτυξης στις ευρωπαϊκές περιφέρειες ε, που θα βοηθήσει τα κράτη-μέλη. Αυτό είναι ένα προευρωπαϊκό ε, και άλλη εργαλείο, ένα εργαλείο, ένα χρηματοδοτικό μέσο, ένα μέσο αλληλεγγύης και τον Ιούλιο όλα αυτά ε, θα μας κάνουν περήφανους ε, γιατί θα μπορούμε να έχουμε καταλήξει σε ένα πολύ σημαντικό πακέτο μαζί με τους υπόλοιπους. Επίσης, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να κάνουμε και κάποια πράγματα για να προωθήσουμε την πολιτική συνοχής. Για παράδειγμα, ε, το θέματα του προϋπολογισμού δεν έχουν ακόμα ξεκαθαριστεί και αυτά επηρεάζουν την πολιτική συνοχής. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν ε, ε, όταν θα κλείσει και το μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό πλαίσιο τι θα κάνουμε, να φτιάξουμε μια καινούρια, μια σύγχρονη πολιτική συνοχής αν δεν έχουμε τον κατάλληλο προϋπολογισμό δεν γίνεται. Νομίζω όμως ότι το Κοινοβούλιο έχει δεσμευτεί γι' αυτό και σε πολλές από τις τροπολογίες αναφέρονται πράγματα που έχουν να κάνουν με τον δημοσιονομικό κανονισμό. Πρέπει να εργαστούμε πάνω σε αυτά, να αλλάξουμε την πρόταση της Κομισιόν, γιατί υπάρχουν κάποιες τροπολογίες που πραγματικά δεν μπορούν να, δεν μπορούμε να τις επεξεργαστούμε ως προς ε, τα αποτελέσματα που θέλουμε. Επίσης, δεν έχουμε ε, νούμερα για τον προϋπολογισμό, κάποιο προϋπολογισμό στην έκθεση. Και οι περισσότερες τροπολογίες παίρνουν κάποια απόσταση από τέτοια νούμερα. Πρέπει σε αυτό το θέμα να βρούμε μια κοινή γραμμή και στις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο θα πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ ε, πώς θα γίνει η διαπραγμάτευση παράλληλα με την αυτήν για το μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό σχεδιασμό. Επίσης, συμφωνήσαμε ότι θα πρέπει να γίνουν και κάποιοι ε, συμβιβασμοί ε, σε κάθε άρθρο και σε κάθε αιτιολογική σκέψη υπάρχουν κάποιοι συμβιβασμοί. Προτείνω όμως στην ψηφοφορία, όταν έχουμε συμβιβαστικές τροπολογίες, να τις έχουμε ως πακέτο. Ας πούμε για το άρθρο 14 να μην έχουμε μία συμβιβαστική τροπολογία με 10 διαφορετικά κομμάτια, να πάει σαν πακέτο, έτσι ώστε η συνένεση που θα προσπαθήσουμε να βρούμε μεταξύ των διαφόρων τροπολογιών και πολιτικών ομάδων να γίνει πιο εύκολη και γι' αυτό το λόγο ζητώ από την Επιτροπή να είναι συνεπής ε, ως προς τον τρόπο που θα ψηφίσει σε αυτές τις ε, συμβαστικές τροπολογίες. Με την πρώτη εξέταση, αν έχουμε ένα άρθρο με πάνω από 200 τροπολογίες, καλό θα ήταν να το συνοψίσουμε σε μία, σε μία συμβιβαστική τροπολογία για να βρούμε έναν λογικό συμβιβασμό. Πιστεύω ότι θα το καταφέρουμε. Ε, φυσικά έχουμε και τροπολογίες οι οποίες είναι δύσκολες ε, ως προς την επεξεργασία τους. Ε, το θέμα του εις διευκόλυνσης Connecting Europe, συνδέοντας την Ευρώπη. Το θέμα των τροφίμων, τροφίμων για τους πτωχούς, το θέμα του «Capping» Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά και πολιτικά και για μας προσωπικά. Πρέπει λοιπόν να δούμε πώς θα τα βάλουμε όλα στο ίδιο καλάθι. Νομίζω λοιπόν ότι έχουμε προχωρήσει αρκετά καλά την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε συνομιλίες και με τους σκιώδεις εισηγητές και την εβδομάδα του Στρασβούργου μαζί με τους σκιώδεις και στις ομάδες εργασίες των ομάδων ε, θα μπορέσουμε να συζητήσουμε τις συμβαστικές τροπολογίες και πιστεύω ότι την Παρασκευή πριν από το Στρασβούργο θα τις έχουμε στα αγγλικά για να μπορέσετε να δείτε και να έχετε γύρω στη μία εβδομάδα χρόνο για να δείτε που είναι τα προβλήματα. Να σας θυμίσω για άλλη μια φορά ότι στις ε, διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο και με την Κομισιόν θα είμαστε επιτυχείς μόνο στο να έχουμε έναν κατάλληλο προϋπολογισμό μόνο αν έχουμε μία έξυπνη προσέγγιση για μεταρρύθμιση της ε, πολιτικής συνοχής. Να είμαστε φίλοι της συνοχής αλλά και των καλύτερων δαπανών. Οι, οι θέσεις θα πρέπει να είναι κοινέ πριν τη διαπραγμάτευση και αν υπάρχουν και περιφερειακές ευαισθησίες να τις βάλουμε και αυτές μέσα. Τις θέσεις του Συμβουλίου που δεν, δεν πρέπει να τις ε, συζητήσουμε, να μην τις βάζουμε σαν τροπολογίες ε, στο Κοινοβούλιο. Αυτό μειώνει λίγο το φόρτο των τροπολογιών μάλλον σε πολύ μεγάλο βαθμό το μειώνει. Και καλό θα είναι να ενισχύσουμε τις δικές μας θέσεις και να αποφασίσουμε στην Επιτροπή με μεγάλη πλειοψηφία για να μπορούμε να έχουμε μια ισχυρή διαπραγματευτική θέση ε, έναντι του Συμβουλίου αλλά και της Κομισιόν. Αυτό είναι η καλύτερη προσέγγιση για να έχουν επιτυχία οι διαπραγματεύσεις και σίγουρα στο τέλος θα έχουμε και καλό αποτέλεσμα από τις διαπραγματεύσεις. Ε, η Ντανούτα είπε ότι συνεχώς πρέπει να αναφέρουμε τι γίνεται και ενδεχομένως να πρέπει να ψηφίσουμε αν υπάρχει κάποια αλλαγή στην εντολή. Αλλά χαίρομαι ιδιαίτερα για τη συνεργασία σχετικά με τις ε, συμβαστικές τροπολογίες και Ελπίζω ότι θα έχουν και μεγάλη υποστήριξη. Ε, είναι λίγο δύσκολο. Ε, πραγματικά, αν διαβάσετε τις τροπολογίες ε, στη γλώσσα σας, θα μπορέσετε να κάνετε κάποια σχόλια και ίσως να έχουμε και μια κατεύθυνση έτσι για τις συμβαστικές τροπολογίες. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν θες κάτι να προθέσεις, Λόμπερ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, είμαι λίγο μπερδεμένος η Κωνσταντζα πιστεύει ότι ίσω όλα πάνε σαν το πρωτάθλημα του ποδοσφαίρου. Η Ολλανδοί είναι ακόμη μέσα. Αλλά εσείς περάσει το επόμενο παιχνίδι. Μη προχωρήσετε πολύ γρήγορα λοιπόν. Τέλος πάντων, ας σοβαρευτούμε. Κωνσταντζα, ήταν πλήρης εξηγώντα τη θέση μας. Το μόνο που θέλω να υπογραμμίσω είναι ότι μετά από την ε, συζήτηση που είχαμε και αυτή που θα έχουμε τώρα και έχοντας ακούσει την Επιτροπή των Περιφερειών, μπορούμε με όλα αυτά τα στοιχεία να εμπλουτίσουμε την πρώτη πρότασή μας. Δεύτερη παρατήρηση. Ξέρουμε μέχρι πού μπορεί να πάει και το Συμβούλιο. Και παρά το γεγονός ότι είχαμε την εντύπωση ότι δεν επιτρέφει μεγάλη πρόοδος κατά της ε, Δανικής ε, Προεδρίας. Από τη μεριά του Συμβουλίου ακούσαμε να λέγεται ότι όντως είναι διατεθειμένο το Συμβούλιο να ε, διαπαραματευτεί μαζί μας. Εξαιρετικό είναι αυτό. Και ακόμη πιο ενδιαφέρον, επειδή συνομοθετούμε σε αυτά τα θέματα, Αυτό δεν σημαίνει ότι απαραίτητο θα καταλήξουμε σε θετικά και εφόρα αποτελέσματα, αλλά εμεί αυτό θέλουμε να δείξουμε και το είπαμε και την τελευταία φορά. Η πολιτική επενδύσεων θα πρέπει να επιτρέπει να έχουμε ανάπτυξη στις διάφορες περιοχές, συνεκτικότητα νέες θέσεις απασχόλησης και ανάπτυξη και πιο πράσινη και συμπεριληπτική Ευρώπη στα πλαίσια των στόχων του 2020. Θα πρέπει λοιπόν στα πλαίσια αυτή της εντολής, όπως είπαμε και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και όλα αυτά, να τα προλάβουμε για να τα ψηφίσουμε τον Ιούλιο. Αν δεν κάνω λάθος, Όλα αυτά μπορούμε να τα διαπραγματευτούμε. Κάποιοι συνάδελφοι όμως από άλλες επιτροπές λέγουν ότι θα πρέπει να είναι πρώτα απ' όλα σαφές πόσα χρήματα θα έχουμε και μετά θα δούμε ε, τι θα γίνει με, τους κανονισμό, με τον κανονισμό. Εμείς όμως τα βλέπουμε διαφορετικά. Θέλουμε να έχουμε μέχρι το τέλος της συζήτησης μία ε, προσέγγιση για η φορεία. Η θέση μας ξέρετε. Είναι αυτή που εξηγήσαμε και στις προηγούμενες συζητήσεις. Και ως συζητητές θέλουμε να εμπλουτιστεί η νομοθεσία για την επόμενη περίοδο. Και αυτό θέλουμε να επιτύχουμε την διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Την επόμενη εβδομάδα θα λάβει χώρα και η διάσκεψη της Συνόδου Κορυφής. Δεν ξέρουμε ότι υπάρχει στα διάφορα κουτάκια. Η Επιτροπή την τελευταία φορά δεν υπάρχει καμία ρύθμιση μέχρι τώρα ε, και τίποτα τότε τελεσμένο με το Συμβούλιο. Και το Συμβούλιο μας λέει, ας κάτσουμε μαζί να το διαπραγματευτούμε. Και κάθε δύο εβδομάδες συναντιέται η αντιπροσωπεία μας με άτομα από το Συμβούλιο. Τη στιγμή που διερχόμαστε όλοι μία κρίση και όλοι διαρωτώμεθα τι καλές επενδύσεις πρέπει να γίνουν, νάτες οι καλές επενδύσεις. Και πρέπει να το πολεμήσουμε αυτό και θα το καταλάβουν οι πολίτες. Και πρέπει να μπορέσουμε να επηρεάσουμε τα πράγματα στη συζήτηση. Εγώ είμαι μέλος και της Ήτρε και στα πλαίσια του προγράμματος Horizon 2020 συζητώνται όλα αυτά τα πράγματα. Όλοι έχουν τα μάτια στραμμένα και στο χρήμα βεβαίως, αλλά και στην συνοχή. Όλοι θέλουν με τη βοήθεια των διαφόρων ταμείων να υπάρξει ανάπτυξη σε αυτή την Ευρώπη που θέλουμε. Και νομίζω ότι αυτό θα επηρεάσει και τη θέση μας και στα πλαίσια της συζήτησης των πολιετούς προγράμματος. Δεν ξέρω αν ε, μακρηγόρησα μετά από αυτά τα οποία είπε η Κωνσταντζα. Ε, δεν θέλω να σε παρηγορήσω, αλλά αυτά που είπες πραγματικά ήταν πολύ σημαντικά. Και όπως είπες, αυτή η πολιτική μπορεί να γίνει σλόγγαν, όπως είπες. Αυτή η πολιτική είναι το σχέδιο επενδύσεων για την Ευρώπη. Τώρα, ε, περνώ στους σκιώδεις. Inverse goes money. Εγώ σκιώδης θα πρέπει να είμαι πιο σύντομος. Ίσως, ε, ναι, είμαι και πιο προκλητικός αυτά τα οποία θα πω πολύ δύσκολο είναι να ευρεθούν ε, ε, ε, συμβαστικές λύσεις. Έχω την εντύπωση ότι και οι, από τη μεριά της Κομισιές θεωρήθηκαν και επαναστατικές προτάσεις των συντονιστών. να μην έχουμε τις επιδόσεις. Εξάντε να έχουμε μια πολιτική ε, σε σχέση με την συνοχή. Ανάθεση των κονδυλίων καταρχάς. Και σήμερα έχω την εντύπωση ότι τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά από ό,τι στην αρχή. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να επιτύχουμε συνέργεια μεταξύ των εθνικών και κοινοτικών συμφερόντων. Θα πρέπει βεβαίως, αν παρακολουθήσουμε τι κάνει κάθε χώρα, κάθε βουλευτή σε κάθε περιοχή, μπορούμε να ακολουθήσουμε κι εμείς να κάνουμε κάτι συνεκτικό με αυτό που γίνεται σε εθνικό επίπεδο. Τι μου έρχεται τώρα κατά νου. Εκεί που θα, πρέπει να καταλήξουμε σε κοινή θέση. Δεν ξέρω πώς θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή, αλλά υπάρχουν ομάδες που κάνουν επαναστατικές ε, προτάσεις. Πρώτα απ' όλα, κάποιοι προτείνουν τρίων ε, ειδών περιοχές να τις διαγράψουμε. Άλλοι να αλλάξουν οι, κάτι, μεταβατικές περίοδο. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να είμαστε ενωμένοι, να μην χωριστούμε στην πληροφορία για αυτά τα θέματα. Δεύτερον, και για τα νέα ταμεία υπάρχουν ε, επαναστατικές προτάσεις. Μακροπεριφερειακά ταμεία, αυτά θα αλλάξουν ε, ε, συγγνώμη, μακροοικονομικές ε, περιοχές έχουμε, αλλά κάποιοι μίλησαν για μακροοικονομικά ταμεία, για μακροοικονομική χρηματοδότηση. Η Κομισιό είπε με τα χρήματα που έχετε κάνετε πολιτική, αλλά μην ζητάτε καινούρια κονδύλια. Αλλά αυτοί που κάνουν τις προτάσεις θέλουν τα χρήματα να πάνε εκεί που πιστεύουν ότι να πάμε. Και εδώ δεν θα, θα πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Επίσης, αυτό το πρόγραμμα, το Connecting ε, Europe, συνδέοντας στην Ευρώπη, είναι κάτι το επίσης μπορεί να χωρίσει κάποιους. Θα πρέπει να δούμε στις μεταφορές. Τι έγινε. Εγώ συνάντησα τον Επίτροπο Κάλλας και θα δοθούν 10 εκατομμύρια όπως είχαν προβλεφθεί για αυτά τα σχέδια μεταφορών τα οποία ήταν πολύ καλά εντός χωρών και πολύ κακά μεταξύ χωρών. Ίσως γι' αυτό θα πω το εξής. Στις χώρες της ε, ε συνοχής δούλεψαν σωστά τα πράγματα. Ο κύριος Μποστινάρου κάτι είπε. Και απήντησε ο, ο Κάλλας ότι εγώ θα δώσω 10 δις για τέτοιου σχέδια. Τι γίνεται αν ε, αλλάξουν ε, οι χώρες αναδύο για τις οποίες θα δοθούν τα κονδύλια για να γίνουν κάποια σχέδια και κάποια προγράμματα. Αν πάντα αναδύο είναι στην συνοχή. Τέλος πάντων, θα πρέπει να βρούμε κάποιες ε, συμβαστικές λύσεις. Επίσης, υπάρχουν κάποιοι με μεγάλες χώρες που έχουν πάρα πολύ μεγάλες περιοχές και εγώ δεν καταλαβαίνω, εγώ είμαι από μικρή χώρα με μικρές περιοχές. Εάν γίνουν πάρα πολλές προτάσεις, είναι εντελώς διαφορετική η προσέγγιση παρά εάν έχετε πολύ μικρές ε, ε, περιοχές. Ε, η Κομισιόν τι θα κάνει, θα κατακαιρματίσει τη δράση και θα μιλάει με τους μικρότερους. Επίσης πρέπει να δούμε τι γίνεται σε επίπεδο ε, ερετών. Υπάρχουν σε κάποιες περιοχές ε, οι ερετοί οι οποίοι κάνουν αυτή την πολιτική της περιφερειακής ανάπτυξης, άλλες όμως υπάρχουν μόνο μικρές ομάδες. Τώρα, στη σχέση με το χρήμα. Δεν ήμουν εδώ στην αρχή, ήμουν στην Επιτροπή Προϋπολογισμών και σήμερα ψηφίσαμε τη γνωμοδότηση για τον κανονισμό, για το Ταμείο Συνοχής, για την εδαφική ε, συνεργασία, για το Κοινωνικό Ταμείο. Αυτό το οποίο είναι καλό είναι ότι ανασχέδιο υπάρχουν μόνο 20 προτάσεις, ούτε 100 ούτε 1000. Δεν είναι τόσο επαναστατιστικές, αλλά κάτι είναι πολύ σοβαρό είναι μία γενική πρόταση που δεν νομίζω ότι θα υποστηριχτεί αργότερα. Είναι ερώτηση προς την Κομισιό ή στο Συμβούλιο, ώστε τα χρήματα για την συνοχή να είναι 5,1% λιγότερα αλλά ακόμη και αν ήταν 5,1% πάνω όπως ψηφίσαμε στην ΣΟΥΡ δεν θα επαρκούσαν. Και το θέμα σε αυτή την πρόταση είναι το εξής. Ποια είναι η απάντηση στο ερώτημα ποιες είναι οι πραγματικές περικοπές. Τίποτα άλλο δεν ήταν επαναστατικό στην Επιτροπή ε, Προϋπολογισμών. Και από ό,τι καταλαβαίνω, θα πρέπει να μπορέσουμε να αναπροσαρμόσουμε τις συνενετικές μας θέσεις και να μην χωριστούμε σε... και να μείνουμε στις θέσεις μας. Να μην αρχίσουμε να λέμε α, πιο προηγμένη περιοχή, λιγότερο προηγμένη, σε μεταβατική περίοδο, γιατί αν χωριστούμε στην ψηφοφορία δεν θα επιτύχουμε τίποτε. Τέλος πάντων, εγώ σας τα από αυτά είναι προσπαθήσω να σας βοηθήσω να διαμορφώσετε άποψη. Ευχαριστώ. Παρακαλώ να είναι πολύ σύντομοι οι επόμενοι ομιλητές, γιατί για το θέμα αυτό έχουμε πολύ λίγο χρόνο, μόνο μισό ώρα. Ο κύριος Γκλάσερ. Κυρίες και κύριοι, θα είμαι πολύ σύντομος. Εγώ εκτιμώ το πολύπλοκο χαρακτήρα του προβλήματος πρέπει να αντιμετωπίσουμε και γι' αυτό και βασίζομαι στις πρώτες συμβιβαστικές προτάσεις τις οποίες ε, περιμένω και ε, φυσικά θα τη συζητήσουμε. Εμπιστεύομαι απολύτως τους συνεισηγητές. Ε, θα μας ενημερώσουν αν υπάρξουν δυσκολίες στις διαπραγματεύσεις, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, αν θέλουμε όντως να είμαστε ενωμένοι ως Επιτροπή και ως Κοινοβούλιο. Είναι ο μόνος τρόπος ε, να, μπορέσει να, μπορέσουμε να πιέσουμε την Κομισιόν να κινηθεί εκεί όπου χρειάζεται να δεχτεί τις προτάσεις μας. Πιστεύω πως θα πρέπει να βρούμε λοιπόν αυτήν ε, την ε, δυνατότητα για άμεση συνεργασία και όχι να μείνουμε στα μεμονωμένα κομμάτια που πρέπει πάντοτε να αναζητούμε τις συμβιβαστικές και να πείσουμε την Κομισιόν ότι πρέπει να κινηθεί και εκείνη από την αρχική της θέση. Δεν είναι μόνο μερής προσπάθεια από τη δική μας πλευρά. Προσβλέπω στις διαπραγματεύσεις και στις συμβιβαστικές. Ευχαριστώ. Κύρια Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα ήθελα καταρχήν να χαιρετήσω τη σημαντική εργασία που έκαναν οι δύο εισηγητές για τον κανονισμό που σίγουρα είναι ένας από τους πιο σημαντικούς που πέρασαν κατά τη διάρκεια αυτής της θητείας. Ε, γενικά είμαστε ικανοποιημένοι ε, γιατί διαγράφεται συνένεση για διάφορα θέματα που θεωρούμε πως είναι πολύ σημαντικά και περιμένουμε τώρα να δούμε τις συμβιβαστικές ε, λύσεις γιατί σήμερα είναι δύσκολο <laughs> να εκφραστεί κανείς για τις 2.000 ε, τροπολογίες. Εγώ θα κάνω κάποιες γενικές φύσεις παρατηρήσεις για τα σημεία που κατά τη γνώμη μου είναι τα πιο κέρια. Πιστεύω πως υπάρχουν δύο στοιχεία τα οποία θα βαρύνουν στις διαπραγματεύσεις που θα ακολουθήσουν, που είναι και που μάλλον διέπουν τις ε, γενικούς προσανατολισμούς πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταρχήν μείωση των δημοσίων δαπανών και από την άλλη πλευρά αμφισβήτηση της δημοσιονομικής κυριαρχίας των κρατών που εκφράζεται μέσα σε αυτόν τον κανονισμό από τους μακροοικονομικούς όρους τους οποίους εμείς αρνούμεθα. Είναι ένα κεντρικό ζήτημα για την ομάδα μας και εκτιμώ πως σε, αυτή την, σε αυτό το θέμα της, ε, των ε, μακροόρων είναι προβληματικό είναι προβληματικό και όσον αφορά τις ευθύνες που θα βαρύνουν τις περιφέρειες, ευθύνες που δεν είναι δικές τους. Επίσης, σε συντομία, θα ήθελα να αναφέρω το θέμα των ε, εξάντε όρων ε, εις βάθος δουλειά θα πρέπει να γίνει για να επαληθεύσουμε μέσα στα παραρτήματα ε, εδάφιο προς εδάφιο πως τα όσα ορίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι καταχρηστικά. Δύο λόγια επίσης για τις νέες κατηγορίες περιφερειών. Περιφέρειες ε, σε μετάβαση. Στην ομάδα μας είμαστε υπέρ της διατήρησης αυτής της νέας κατηγορίας και θα αντιταχθούμε, δεν φαντάζομαι πως θα σε εκπλήσει αυτό, στις προτάσεις και στις τροπολογίες που θέλουν να καταργήσουν αυτή την κατηγορία κατηγορία τριών διαφορετικών κατηγοριών περιφερειών θεωρούμε πως είναι δίκαιη και ισότιμη λύση και αυτό μάλιστα γιατί οι περιφέρειες που βγαίνουν από τον πρώην στόχο 1 θα έχουν ένα μίνιμουμ 60%, 70% ε, συγγνώμη, των κονδυλίων που εγγυημένο ε, των κονδυλίων που είχαν το η περίοδο 2007 μέχρι 2013. Ένα θέμα στο οποίο θέλω να επιστήσω όμως την προσοχή σας είναι το θέμα των ιδιαίτερα απομακρυσμένων περιοχών περιφερειών. Το έχουμε συζητήσει. Είναι και η Αυστρία και η Σουηδία ε, μέσα σε αυτές τις ε, περιοχές. Έχουμε υποβάλει σχετική τροπολογία και θα την υπερασπιστούμε και προτείνουμε το κονδύλι να μην μειωθεί. Η Επιτροπή μας μάλλον η γνώμη της Επιτροπής μας αναμένεται με ανυπομονησία από όλες τις ε, ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιοχές. Παρά λοιπόν αυτές τις επιφυλάξεις ε, θα ήθελα να σας συγχαρώ για το κλίμα που επικρατεί στην Επιτροπή μας για την αναζήτηση συνένεσης ε, για τα πιο σημαντικά θέματα. Σας ευχαριστώ. Ο Ευχαριστώ ε, και Πρόεδρε που μου δίνετε την ευκαιρία να συμβάλλω και εγώ σε αυτή τη συζήτηση. Καταρχήν να συγχαρώ τους δύο συνεισηγητές για το σχέδιο έκθεσης και για τις ε, τροπολογίες. Πολύ καλή βάση για την περαιτέρω εργασία μας για το νομοθετικό πακέτο περί πολιτικής συνοχής. Ε, έχουμε τη θεματική συγκέντρωση. Καταρχήν πιστεύω πως η νέα προγραμματική περίοδος θα πρέπει ε, για την συνοχή, πολιτική συνοχή θα πρέπει να είναι πιο στοχοθετημένη, φιλική προς το δικαιούχο και, αποδοτική. Άρα λοιπόν η, ευελιξία είναι απαραίτητη γιατί θα επιτρέψει τη θεματική, το μέσο μάλλον θεματικής συγκέντρωσης να αντικατοπτρίζει τις εξελίξεις στις περιφέρειες και να επιτύχει τους στόχους της. Στους ε, συναδέλφους που πιστεύουν ότι μπορεί να είμαστε επαναστατικοί. Δεν είναι κακό αυτό. Μερικές φορές χρειάζεται και γι' αυτό και στηρίζω την πρόταση της Κομισιόν για τα αποθεματικά απόδοσης. Αυτό νομίζω ε, είναι αμφισβητήσιμο για το κατά πόσο τελικά θα ε, ωφελήσει την πιο αποδοτική περιοχή. Ε, θα άλλο σημείο που αφορά τον ΦΠΑ ε, υποστηρίζω την πρόταση του εισηγητή ώστε να αφαιρέσει την ε, διάταξη που αφορά τον ΦΠΑ που δεν είναι εισφρακτέως υπό την εθνική νομοθεσία ΦΠΑ και επίσης υπό την Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία η συγχρηματοδότηση θα πρέπει να ανέρχεται στο 85% αντί για το 75%. Έτσι τα κράτη-μέλη θα είναι πιο φιλόδοξα και έτσι θα αυξηθεί και ε, το ποσοστό απορρόφησης. Κάτι που επίσης αναφέρθηκε από κάποιους προηγούμενους ομιλητές είναι η εμπλοκή των ενδιαφερομένων φορέων στον φάση προγραμματισμού. Είναι σημαντική, ίσως όχι με ομάδες δράσης, αλλά εν πάση περιπτώσει δικαιούχοι ενδιαφερόμενοι εμπλεκόμενοι φορείς και έχω καταθέσει σχετικές τροπολογίες, αν και η πρόταση της Κομισιόν καλύπτει καλά και αυτό το σημείο. Σας ευχαριστώ πολύ και θα αναμένω με ανυπομονησία τις συμβιβαστικές. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα, συνάδελφε, να κλείσω τον κατάλογο. Έχουμε την κυρία Μανέσκου, Πίπερ, Τόγερ. το Mr. Uh, Madame Smolkova. Μπορούμε να ακούσουμε την κυρία Σμόλκοβα ε, επίσης. Ε, όχι πάνω από τρία λεπτά όμως ο καθένας. Είτε θα πάρετε δύο λεπτά και θα ακούσω περισσότερους, είτε το άλλο. Ε, Αύριο έχουμε άλλη μια ώρα. Ό,τι θέλετε. Αποφασίστε. Κλείνω με την κυρία Σμόλκοβα. Δεν μπορούμε να έχουμε την κυρία Σμόλκοβα γιατί έχουμε το σκιώδη συγητή. Εκεί σταματάμε και τώρα η κυρία Σρέτερ ως σκιώδης. Εκτός από τον κύριο Αλφόνση. αντί, αντί του κυρίου Αλφόνση μάλλον και αύριο έχουμε άλλη μία ώρα. Ελίζαμπετ, έχεις το λόγο. Υπέροχα. Ευχαριστώ. Καταρχάς βρισκόμαστε στη φάση των διαπραγματεύσεων. Γι' αυτό το λόγο και εγώ ε, ταξιδεύω πολύ. Παραδόθε. Είναι σημαντικό να έχουμε μία συμφωνία. Να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Καταρχάς, θεωρώ ότι η ιδέα με το κοινό στρατηγικό πλαίσιο, να πω ειλικρινά, αποδέχομαι τη δουλειά του εισηγητή σε αυτό το θέμα, αλλά μπορώ να πω ότι δεν τα έχουμε καταφέρει να βγάλουμε ένα καλό σχέδιο όταν ε, βλέπει κανείς πόσα πράγματα μπήκαν μέσα. Επίσης, ε, ομολογώ ότι και εγώ δεν κατάφερα να πείσω για ένα σχέδιο τροποποίησης. Γιατί όταν κοιτάει κανείς, ε, βλέπει ότι κάθε λέξη συμβάλλει την ίδια εικόνα. Από τη στιγμή που έχουμε ε, αν είχαμε ένα καλύτερο ε, κείμενο θα περιορίζαμε τα κράτη-μέλη ως προς τη χρήση των διορθωτικών ταμείων και αυτό δεν θα έπρεπε να το κάνουμε. Είναι μια κακή εικόνα του Κοινοβουλίου το να συμβάλλει σε κάτι τέτοιο, το να βοηθάμε ε, στην απλούστευση είναι το σωστό, ανταυτού εμείς ε, ε, περιπλέκουμε. Τι σημαίνει σκέφτηκα για τα κράτη-μέλη να έχουμε αυτές τις προϋποθέσεις που βάζουμε με τις τροπολογίες είτε με τις δικές μου είτε με τον ε, όταν προσπαθούν να κάνουν ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα. Εγώ θα είπα ότι η ίδια δεν θα ήθελα να έχω μια τέτοια διαχείριση να κάνω. Πρέπει λοιπόν σε αυτό το επίπεδο να δούμε τι θα γίνει με το κοινό στρατηγικό πλαίσιο. Να έχουμε ένα έγγραφο το οποίο θα μας δίνει καθοδήγηση για το πώς κάνει κανείς κάτι και αυτό θα το αφήσουμε στην Κομισιόν. Γιατί εκεί μπορούν πολλοί να εξετάσουν και να δουν πώς αυτό θα είναι βοήθεια για τα κράτη-μέλη και να μην έχουμε ε, κανόνες οι οποίοι θα είναι σε επίπεδο κανονισμού πολύ καλοί, αλλά στην πραγματικότητα δεν θα λειτουργούν και θα πρέπει να γυρίσουν από εδώ και από εκεί για να τα βγάλουν πέρα. Άρα, νομίζω ότι θα πρέπει από κοινού να σκεφτούμε και ίσως να αλλάξουμε το κείμενο ή να κρατήσουμε κάποια στοιχεία αλλά να μην το κάνουμε τόσο ε, αυστηρό σε επίπεδο κανονισμού, να το κατεβάσουμε λίγο. Νομίζω ότι δεν μπορούμε να ζητάμε από τους άλλους να κάνουν μια διαχείριση με βάση αυτές τους όρους και τις προϋποθέσεις και απλά να ε, ψώνουμε τη σημαία των δημοκρατικών δικαιωμάτων. Νομίζω ότι πρέπει να βρούμε μια ισορροπία ανάμεσα στην διαφύλαξη των δημοκρατικών δικαιωμάτων και στην ύπαρξη ενός λογικού κανονισμού, ο θα μπορέσει να εφαρμοστεί. Uh, Ευχαριστούμε, κυρία Μανέσκου. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ήθελα πρώτα απ' όλα να συγχαρώ τους δύο συνεισηγητές για την εργασία που επιτέλωσαν. Μεγάλος φόρτος και έκαναν πολύ καλή δουλειά και με τις τροπολογίες. Είμαι σίγουρη θα μπορέσουν να επιλέξουν τις καλύτερες δυνατές συμβιβαστικές ε, τροπολογίες. Νομίζω ότι θα μπορέσουν να γίνουν διάφορες αναπροσαρμογές και οι συγητές και οι συνεισηγητές θα μπορέσουν να κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά για την διαπραγμάτευση. Για αν σκεφτώ κατά πόσον μπορούμε για τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις να τονίσουμε την ε, καινοτομία και την δυνατότητα προσαρμογής γιατί είναι πολύ σημαντικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση νομίζω ότι θα μπορέσουν στα πλαίσια του νέου ε, κανονισμού και στα πλαίσια της πολιτικής συνοχής να συμπεριληφθούν περισσότερες μιμιέ και μικρο Είναι πολύ σημαντικό στο άρθρο 1 να κάνουμε αναφορά στο Small Business Act for Europe, ώστε να μπορέσουμε να λάβουμε υπόψη την επικοινωνία των ΜΜΕ και να κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε να μπορέσουμε να διευκολύνουμε την πρόσβασή τους στις στη μικροχρηματοδότηση. Ένα άλλο σημείο και την άποψή μου είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι αυτό της τεχνικής αρρωγής, το άρθρο 51 που προβλέπει η Κομισιό. Ή οι πολύ πολύπλοκες διαδικασίες ή η έλλειψη επικοινωνίας και ενημέρωσης και συμμετοχής των τοπικών ε, μετεχόντων αποθάρρυναν τις ΜΜΕ από το να συμμετάσχουν σε όλη αυτή τη διαδικασία βοήθειας μέσω των ταμείων. Είδαμε τις ε, εκθέσεις της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είδαμε τις εκθέσεις του Ελεκτικού Συνεδρίου, Είδαμε ποιες είναι οι αδυναμίες, αλλά για να μπορέσουμε να είμαστε συνεκτικοί, θα πρέπει στο άρθρο 51 να προσθέσουμε ότι είναι αναγκαίο να καταρτίζονται και να ενημερώνονται όλοι μας οι εταίροι έτσι όπως προβλέπετε. Η ανάγκη λοιπόν αυτή να έχουν την κατάλληλη κατάρτιση και ενημέρωση οι υπεύθυνοι των διαφόρων προγραμμάτων, ώστε να αποφευχθούν εμπόδια ή σφάλματα τα οποία θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν. Δεδομένου ότι σε παρούσα περίοδο πρόκειται για σημαντικά προσκόμματα. Μία άλλη παρατήρηση αφορά το άρθρο 29, στρατηγική τοπικής ανάπτυξης. Θα πρέπει να αναφερθεί στο άρθρο 5 διορθώνει η συγγετρία. Στο 5 προβλέπονται οι εταίροι και ιδιαιτέρως οι κοινωνικοί εταίροι θα πρέπει να είναι μέλη της Επιτροπής Επιλογής. Διότι αυτή η αρχή της εταιρική σχέσης είναι πολύ σημαντική. Συζητήσαμε διαμαχρόνια και νομίζω ότι εδώ υπάρχει συνένεση. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να αναφέρουμε με απόλυτη σαφήνεια ποιοι είναι οι εταίροι οι οποίοι θα μπορούσαν να τύχουν τεχνικές βοήθειες. Και να πούμε επίσης ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να ζητήσουν από ιδιώτες και από τις τοπικές τους αρχές να εμπλακούν σε όλα αυτά τα σχέδια, τα εταιρικά που συνάπτουν για την ανάπτυξη περιοχής τους. Είδα ότι πολλές τροπολογίες κατατέθηκαν για τα θέματα αυτά, όχι μόνο εκ μέρους του Άλντε, αλλά εκ μέρους και άλλων πολιτικών ομάδων. Γι' αυτό πιστεύω ότι θα μπορέσουν όλες αυτές οι τροπολογίες να αποτελέσουν αντικείμενο συνενετικής τροπολογίας δεδομένου ότι έχει υπάρξει, όπως σας είπα, ε, συμφωνία. κύριος Πίπερ. Ευχαριστώ. Μιλάμε για τη μεγαλύτερη τμήμα του προϋπολογισμού σε επίπεδο ευρωπαϊκό. Και είμαστε σε μια συζήτηση η οποία είναι ήσυχη, ε, αντι, πολύ χωρίς εντάσεις και πραγματικά αυτό δεν το καταλαβαίνω. Ε, δηλαδή ε, πάω σπίτι μου και λέω πού βρίσκομαι. Στις ευρωεκλογές πηγαίνω στους, στην εκλογική μου περιφέρεια και με ρωτάνε πού τι κάνουμε. Ε, ποια είναι η θέση των σοσιαλιστών, των πρασίνων. Το να βρίσκουμε συμβαστικές λύσεις ε, τόσο ήσυχα με ξεπερνά. Το να έχουμε δηλαδή ίδιες θέσεις οι χριστιανοδημοκράτες με τους σοσιαλιστές για το θέμα της ανάπτυξης, δεν ξέρω. Η συζήτηση πραγματικά με ανησυχεί και θα έπρεπε να μας ε, κάνει να έχουμε πιο μεγάλη ένταση. Ας πούμε, η κυρία Κρέλ λέει ότι πρέπει να ψηφίσουμε σε πακέτα για να προχωρήσουμε. Εγώ δεν μπορώ να υποσχεθώ με τις δικές μου τροπολογίες ε, να συμβάλλω σε κάτι τέτοιο, γιατί είναι πράγματα τα οποία θεωρώ βασικά και θεμελιώδη. Πρέπει να τα συζητήσουμε σε βάθος πραγματικά θα έχω και κάποιους συμμάχους σε αυτή τη στρατηγική. Να αναφερθώ σε ένα-δύο σημεία. Πρώτον, το θέμα που ε, ε, έχει να κάνει με την καλύτερη διασύνδεση των ε, διαρθρωτικών ταμείων με τα ευρωπαϊκά δίκτυα και την διευκόλυνση συνδέοντας την Ευρώπη. Θα προσπαθήσουμε να περάσουμε τα χρήματα στην Κομισιόν ε, ώστε να μπορεί ε, στα κράτη-μέλη να γίνεται σωστή χρήση τους. Αυτό δεν το θέλει η Κομισιόν, αλλά πραγματικά νομίζω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ήταν καλό να, υπάρχει, να προωθήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση να υπάρχει μεγαλύτερη ευθύνη από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τη συμβάση εταιρική σχέσης τώρα. Υπάρχει η κατηγορία η μεταβατική, θέλω να τη θίξω λιγάκι. Ε, πάντοτε ελπίζω ότι θα υπάρχει συμβιβασμός. Ξέρουμε ποια είναι η πρόταση της Κομισιόν, θεωρώ ότι δεν είναι σωστή. Το να βρούμε ένα συμβιβασμό, να πούμε εντάξει μια ε, μεταβατική κατηγορία, αλλά να έχουμε ένα ανώτατο όριο ε, σε διάρκεια για την ε, επιχορήγηση των περιφερειών. Εμένα στο, εμάς στο ΕΛ, για μένα στο ΕΛΚ και από τους φιλελεύθερους υπάρχει κάποια υποστήριξη και αυτό ε, ισχύει και για άλλες ομάδες γιατί δεν μπορούμε να βρούμε συμβιβασμό. Με 40 και 50 ε, ψηφοφορίες το να αποφύγουμε να μην βρούμε συμβιβασμό είναι λίγο δύσκολο. Να συνεχίσουμε έτσι. Θα πρέπει να προχωρήσουμε και να προσπαθήσουμε στο τέλος να βρούμε συμβιβασμό. Ε, Ευχαριστούμε, Μίκαλ Τόιρερ. Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να, χρησι... να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία και να πω κάποια πράγματα σχετικά με τον δημοσιονομικό κανονισμό στη συνάδελφο Κρέλ. Είχαμε ε, μία τριμερή συνάντηση στην Επιτροπή Προϋπολογισμού και Ελέγχου του Προϋπολογισμού και νομίζω ότι όλα αυτά ε, έχουν να κάνουν με όλες τις spending committees, της επιτροπές δαπανών. Αυτά που γίνεται στο Συμβούλιο πολλές φορές ε, με κάνουν να σκέφτομαι πολύ. Νούμερο ένα, ε, μιλάμε για νέα χρηματοδοτικά μέσα για τους επικεφαλείς κρατών και κυβερνήσεων Αυτά ε, είναι συγκεκριμένα. Τώρα ε, μιλάμε ε, και υπάρχει μεγάλη ασυμφωνία σχετικά με το αν θα πρέπει να υπάρχουν επιστροφές. Αυτό είναι ένα παράδειγμα. Στο άρθρο... Ε, 56 και 77 υπάρχουν κάποιες τροπολογίες του Κοινοβουλίου υπάρχει τεχνικής, τεχνικός και πολιτικός ε, τρίλογος και η Κορεπέρ και αυτό καταλαβαίνω ότι δεν θα οδηγήσει σε συμφωνία στην πρώτη ανάγνωση. Είναι ένα πρόβλημα λοιπόν να έχουμε τέτοιους τομεακούς κανονισμούς, αλλά σε αυτή τη φάση θα πέσει να μην υποχωρήσουμε, θα πρέπει να μην υποχωρήσουμε και να εξασθενήσουμε τη θέση του Κοινοβουλίου. Ίσως το ένα ή το άλλο θέμα στον κανονισμό, τον περιφερειακό ή του προϋπολογισμού μπορεί να είναι πολύ συγκεκριμένο και ειδικό και ίσως θα μπορούσαμε να το κάνουμε πιο απλό, αλλά υπάρχουν και κάποια άλλα περιφερειακά ζητήματα στα οποία πρέπει να μένουμε σταθεροί. Θα πρέπει να διαφυλάξουμε το δικαίωμα ελέγχου του Κοινοβουλίου, να υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες να υπάρχει ε, μια επιρροή από την Επιτροπή, αλλά να συνδέεται με τους στόχους μας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Να τηρούμε αυτούς τους στόχους, γιατί αλλιώς δεν έχει νόημα. Ακούω, ας πούμε, ότι η Κομισιόν έδωσε, θα δώσει τη δυνατότητα να κάνουμε δημοσιονομικές διορθώσεις. για να έχουμε καλή συνείδηση Ήθελα να φέρω αυτή την πληροφορία στην Επιτροπή γιατί με αυτόν τον τρόπο βλέπουμε ότι προσπαθούν ίσως από το Συμβούλιο να διχάσουν το Κοινοβούλιο με την... να έχουμε άλλες θέσεις από την Επιτροπή ε, Προϋπολογισμού, Ελέγχου του Προϋπολογισμού, Γεωργίας, Ανάπτυξης και καλό θα ήταν να είμαστε μαζί σαν μια γροθιά ώστε να μπορέσουμε να επηρεάσουμε σε αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Γιάνν. Γιάνν Ολμπριχτ. Πρόεδρε. Κάποιες... Κάποιες παρατηρήσεις θέλω να κάνω, κύριε Πρόεδρε. Πρώτο απ' όλα, την αισιόδοξη. Μετά από αυτά είπε ο κύριος Πάιπερ. Εάν μια συμβασμό, συμβασμό. Διαφορετικά δεν είναι συμβασμό. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο συμφωνούμε και αν υπάρχει σε κάτι δεν συμφωνείτε, δεν είναι συμβαστική λύση. Θα το ψηφίσουμε χωριστά. Εάν λοιπόν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, δεν θα το θεωρήσουμε ως συμβαστική λύση, ας το συμφωνήσουμε όμως. Εάν είναι έτσι τα πράγματα, θα, θα κάνω τις εξής παρατηρήσεις. Ακούσαμε από την Επιτροπή Περιφερειών ότι υποστηρίζει τις απόψεις μας ότι ότι θα πρέπει να υπάρχει η απόφαση το παράρτημα του κανονισμού. Στα πλαίσια της συναπόφασης σημαίνει ότι και εμείς θέλουμε και το Συμβούλιο το παράρτημα. Μετά από την πρώτη συνάντηση με τη Δανική Προεδρία Ποια είναι η απόφαση στην οποία καταλήξαμε μαζί με το Συμβούλιο για το παράρτημα. Αν είπανε ναι, προχωρούμε. Αν είπανε όχι, να μην χάνουμε χρόνο και ας το αφήσουμε κατά μέρος. Δεδομένου ότι είναι επίγον θέμα. Δεύτερον, το Connecting Europe Facility. Σε όλες τις τροπολογίες εγώ πρότεινα διαγραφή. Για ποιο λόγο? Διότι, όπως και κάποιοι συνάδελφοι που συνάντησαν τον Επίτροπο Κάλλας, με τον οποίο ο οποίος είχε πάρα πολλές συναντήσεις, εγώ κατάλαβα ότι δεν έχει καμία σχέση το Connecting Europe Facility με την πολιτική συνοχή. Αυτό είναι το μήνυμα που έλαβα από τη συνάντησή μου με τον κύριο Κάλλας. Είπε ότι τα χρήματα θα προσθεθούν, θα, θα φύγουν από το Ταμείο Συνοχής αλλά όταν φύγουν δεν θα είναι δικά του πλέον. Χάνουν αυτό το χαρακτηρισμό. Και το νέο μέσον, το οποίο θα δοθεί σε έναν ειδικό οργανισμό της Ευρώπης, που θα είναι στις Βρυξέλλες. Θα είναι κονδύλια, τα οποία δεν θα δοθούν ούτε αναλλαγικά στα κράτη-μέλη, και θα υπάρξει μειοψηφικός διαγωνισμός για να μπορέσουν να επιλεγούν τα προγράμματα που θα υποβληθούν. Αν λοιπόν έτσι είναι τα πράγματα, γιατί να το έχουμε στον κανονισμό για τα μία συνοχή. Γι' αυτό εγώ δεν επιμένω, απλώς λέγω ότι δεν είναι η θέση τους εγώ. Τώρα, αν ληφθεί αυτή η απόφαση, δεν σωστό να το κρατήσουμε εδώ. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα πρόκειται για κονδύλια του Ταμείου Συνοχής. Και τελευταία παρατήρηση, υποστηρίζω αυτά που είπε ο κύριος Κόβατς για την ε, συνεργασία. Δεν πρέπει εμείς για την χρυσή ε, χρηματοδότηση να κατέβουμε κάτω από το 85. Υπογραμμίσαμε πόσο σημαντικό είναι το θέμα της εδαφικής συνεργασίας. Νομίζω ότι θα πρέπει να επιμείνουμε στο 85 και να μην αλλάξουμε θέση. 85%. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, συγγνώμη, μια στιγμή, μια στιγμή θα σας δώσω το λόγο αν περιμένετε. Ο κύριος Νίλσεν ζήτησε πρώτα απ' όλα το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Εάν μου επιτρέψετε θα μιλήσω σου ειδικά γιατί είναι πιο απλό για μένα. Πρώτα απ' όλα πρέπει να πω ότι με εντυπωσιάζει η εξαιρετική εργασία και η θέση που εξέφρασαν οι συγητές, καθώς και οι προσπάθειες να επιτύχουν ευρεία συνένεση. Διότι είναι σημαντικό, για αυτό το σημαντικό θέμα υπάρξει μεταξύ μας, ε, ε υπάρχουν αποκλίνουσες απόψεις, δεν θα έχουμε ισχυρή διαπραγματική θέση. Δεν μπορούμε να έχουμε συμφωνία για τα πάντα, αλλά θα πρέπει να είμαστε ενωμένοι για τα κυριότερα θέματα. Επίσης, πρέπει να πω ότι όταν οι μεγάλες συμβιβαστικές ε, λύσεις επιτευχθούν για την αρχή της εταιρικής σχέσης, θα μπορέσουμε να καταθέσουμε τροπολογίες, διότι σε περιφερειακό επίπεδο η εταιρική σχέση είναι πάρα πολύ σημαντική, ώστε να υπάρχει δύναμη μεγάλη για να μπορέσει η πολιτική συνοχής να γίνει πράξη. Δεδομένου ότι πρόκειται για πολιτική που βασίζεται σε στρατηγική περιφερειακή στα πλαίσια της, ε, των στόχων του 2020 και έτσι μπορούμε να δημιουργήσουμε με τις δραστηριότητες αυτές ανάπτυξη. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό αυτό το θέμα και δεν θα πρέπει να βρεθούμε σε μια κατάσταση για την οποία κάποιες ε, περιφέρειες ε, χάρη της ευελιξίας δεν θα πάρουν κάποιες ευθύνες. Τις ευθύνες τις παίρνουν οι περιφέρειες και πρέπει να συμμετάσχουν οι πολίτες και οι οργανώσεις πολιτών και οι πάντες όσοι βρίσκονται Ευχαριστώ. Πολύ σύντομη κυρία Σμόκοβα. Ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομη γιατί θα μιλήσω πιο πολύ αύριο. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα καταρχάς να ζητήσω συγγνώμη στους συζητητές που κατέθεσα πολλές ε, τροπολογίες. Νομίζω ότι σε εκείνη τη φάση ήταν πιο εύκολα να γράψω 226 τροπολογίες, αλλά καταφέραμε τελικά να τις ε, κάνουμε 250. Με τη συμφωνία του συντάκτη, του συνσυντάκτη, ε, ε, κρατήσαμε τους μεταφραστές ε, απασχολημένους. Να πω τώρα γιατί καταθέσαμε όλες αυτές τις τροπολογίες. Είναι ένα κείμενο που το έχω και στα αγγλικά και δεν θέλω να θα δαπανίσω τώρα το χρόνο σας. Απλά να πω ότι Συμφωνώ με τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιφοριών. Ήδη αναφέρθηκε ότι δεν υπήρχε μηχανισμός υπερεθνικής συνεργασίας, όπως ονομάζεται. Ήταν επαναστατικές ε, οι προτάσεις, αλλά νομίζω ότι είμαστε σε περίοδο επαναστάσεων, οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Από την Κομισιόν, Νίκολας Μάρτιν, ε, ε, υποδιευθυντής, υπογενικός διευθυντής. A few, uh, uh, γενικός Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η Κομισιόν δεν είχε τη δυνατότητα ως τώρα να χωνέψει τον τεράστιο ρυθμό τροπολογιών που έχουν κατατεθεί. Αυτό που θα έλεγα είναι ότι καλωσορίζουμε αυτό το μέγεθος ε, των τροπολογιών. Δεν θεωρούμε ότι η πρόταση της Κομισιόν δεν έχει ποιότητα και γι' αυτό χρειάζεται τροπολογίες. Απλώς ε, αντικατοπτρίζει αυτό την σημασία του πακέτου και πραγματικά ε, μας δίνεται έτσι η δυνατότητα να το βελτιώσουμε και να έχουμε νομοθεσία υψηλής ποιότητας που θα καλύπτει όλα τα θέματα. Να πω κάτι για το κοινό ε, στρατηγικό πλαίσιο, συγκεκριμένα για την ε, Επιτροπή των Περιφερειών, υπάρχει ε, ένα στοιχείο που μπορεί να μας βοηθήσει. Είναι οι key actions, οι βασικές δράσεις. κ. το ανέφερε. Στο σημείο 13 της έκθεσης θα δείτε τη διατύπωση. Δείχνει την άποψη της Κομισιόν σχετικά με αυτές τις σημαντικές και βασικές δράσεις αναφέρεται ξεκάθαρα ότι δεν είναι υποχρεωτικές δράσεις, αλλά είναι παρεμβάσεις προτεραιότητας για να μπορέσουμε να επιτύχουμε την καλύτερη δυνατή προστιθέμενη αξία. Αυτός είναι ένας ε, τρόπος διατύπωσης και πρέπει να τον έχουμε υπόψη μας ε, στην περαιτέρω δουλειά που γίνεται επί ε, του στρατηγικού πλαισίου. Τώρα, η η θέση της Κομισιόν που εκφράστηκε από τον Επίτροπο σε σχέση με το κοινοστατικό πλαίσιο έχει κάποια στοιχεία που αναφέρονται στο σχέδιο εργασίας της Κομισιόν τα οποία μπορούν να συμπεριληφθούν ως παράδειγμα στον κανονισμό κοινών διατάξεων και μπορεί η Κομισιόν να συνεργαστεί με τον εισηγητή για να βρουν αυτά τα σημεία. Επίσης, η προσέγγιση συμπληρώνεται με τις πράξεις κατεξουσιοδότηση που ε, έτσι ε, θα μας δώσουν και μια βάση για διάφορα στοιχεία που έχουν να κάνουν με τους μηχανισμούς συντονισμού και για τα στοιχεία πολιτικής που μπορούν να πάνε στο παράρτημα και πιο ε, λεπτομερή στοιχεία που σχετίζονται με τις βασικές δράσεις και θα είναι και τα στοιχεία που στην πράξη θα δώσουν μια εδαφική ας πούμε, διάσταση που μπορεί να μπει στις ε, πράξεις κατά εξουσιοδότηση. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό σε επίπεδο διατύπωσης γιατί από τη μία βλέπουμε και τα δύο αυτά στοιχεία και το ε, παράρτημα και της ε, κατεξουσιοδότηση πράξης που είναι δεσμευτικά νομικά έγγραφα αλλά δεν θέλουμε με αυτόν τον τρόπο να περιορίσουμε στις εταιρικέ συμβάσεις ε, και προγράμματα, αλλά να δώσουμε μια ευέλικτη καθοδήγηση που θα πρέπει να διατυπωθεί, διατυπωθεί με τον κατάλληλο τρόπο, δεδομένου ότι είναι νομική πράξη. Είναι ένας ε, τομέας αυτός ε, όπου μπορούμε να δώσουμε κάποιες, κάποια καθοδήγηση, κάποιο προσανατολισμό προς το πώς μπορεί να επιτευχθεί κάτι τέτοιο αυτό που θα πρέπει να περιλαμβάνουν οι τροπολογίες θα πρέπει να είναι μια διάταξη που θα προβλέπει τις πράξεις κατεξουσιοδότηση. Η άποψη της Κομισιόν λέει ότι οποιαδήποτε τροποποίηση του παράρτημα θα πρέπει να μπορεί να γίνεται και μέσω από πράξη κατεξουσιοδότηση από τον Κομισιόν αν χρειάζεται αναθεώρηση του παραρτήματος. Ένα τελευταίο σύντομο σχόλιο γιατί δεν έχουμε χρόνο. Μια γενική σκέψη για τη διατύπωση των τροπολογιών. Νομίζω ότι από την πλευρά τη Κομισιόν υπήρχε αυτή η ανησυχία ότι σε κάποιες περιπτώσεις οι προτινόμενε τροπολογίες βασίζονται σε κάποιες περιπτώσεις σε, μια μη σωστή ανάγνωση του κειμένου. Ένα παράδειγμα είναι ε, το αποθυματικό με βάση ε, την απόδοση, τις επιδόσεις. και, πριν από λίγο έγινε μια αναφορά γι' αυτό ε, και αναφέρθηκε ότι σχετίζεται με τις ε, περιοχές που έχουν την καλύτερη απόδοση. Αλλά δεν ισχύει αυτό, δεν έχει να κάνει με τις ε, περιοχές που έχουν την καλύτερη απόδοση. Είναι τα προγράμματα που πληρούν τα συγκρίσιμα κριτήρια που έχουν τεθεί για αυτά τα προγράμματα. Μεταξύ προγραμμάτων, μεταξύ περιφερειών, μεταξύ κρατών μελών, ε, μεταξύ αυτών είναι η σύγκριση. Ε, έχει να κάνει με... Ε, δεν, είναι, δεν είναι μάλλον μεταξύ αυτών η σύγκριση, είναι καθαρά για το αν ένα συγκεκριμένο έργο πληρεί αυτές τις προϋποθέσεις. Οπότε να κοιτάτε πάντοτε οι τροπολογίες να βασίζονται σε σωστή κατανόηση του κειμένου. Τις επόμενες ημέρες η Επιτροπή με τον εισηγητή θα συνεργαστούν με, εμά ώστε να τους βοηθήσουμε κατά την εξέταση των τροπολογιών. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ Νίκολα. Ε, από ό,τι κατάλαβα αύριο θα συνεχίσουμε τη συζήτηση. Αύριο στις 11.30 έχουμε άλλη μια ώρα για να συζητήσουμε το γενικό κανονισμό. Τώρα δίνω το λόγο στον Μάρκο Πίπερ για να συζητήσουμε το θέμα της ε, νομοδότησης για το είναι διευκόλυνση συνδέοντας την Ευρώπη που έχει συντάξει ο Μαρκούς Πίπερ. Ja, vielen Dank. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ως Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης έχουμε την δυνατότητα να πούμε κάτι στην Επιτροπή Μεταφορών σχετικά με την διευκόλυνση συνδέοντα στην Ευρώπη. Νομίζω ότι περισσότεροι συνάδελφοι ξέρουν περί τίνο πρόκειται. Γι' αυτό θα πω σύντομα δύο-τρία. δυο αλλαγές που ε, θα, ήταν, θα άξιζαν τον κόπο να γίνουν ε, από την δική μας πλευρά. Καταρχάς, ε, σε επίπεδο βάσης, θεωρώ ότι η διευκόλυνση συνδέοντας στην Ευρώπη είναι ένα εξαίρετο εργαλείο. Εμείς ως Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης δεν θα πρέπει να φοβόμαστε ότι θα, μας, θα, θα φύγουν χρήματα. Αυτό το μέσο θα οδηγήσει ώστε να γίνουν ε, πιο ε, ισχυρές και να αναπτυχθούν μαζί οι περιφέρειες της Ευρώπης. Για να έχουμε ε, μια βελτίωση των ε, συνδέσεων μεταφορών στην Ευρώπη και οι περιφερειακές περιοχές, αυτές που είναι μειονεκτούσες, να μπορούν να συνδεθούν με τα διαευρωπαϊκά δίκτυα και να επωφεληθούν η κάθε μία από αυτές από αυτό το εργαλείο το συνδέοντας στην Ευρώπη. Ε, σε επίπεδο ανταγωνισμού είναι πολύ καλό. Υπάρχει μια αποτελεσματική χρήση ε, χρημάτων. Τα 10 ε, δις ε, θα πρέπει αναλογικά να διανεμηθούν στους κατοίκους. Αυτό από την άλλη δεν ξέρω αν είναι τόσο... Θεωρώ ότι είναι καλό. Από την άλλη να πω ότι είναι επίγον η διευκόλυνση συνδέοντας στην Ευρώπη να συνδεθεί πιο στενά με την πολιτική συνοχής και τις διαρθρωτικές πολιτικές, έτσι ώστε να συμπληρώνει μία την άλλη. Να μην είναι ένα παράλληλο εργαλείο, αλλά με τα κρατημέλη, με τις περιφέρειες να υπάρχει εφαρμογή. Ε, για να έχει απόλυτο δίκιο σε αυτό. Αν δεν υπάρχει συνεργασία δεν θα προχωρήσουμε πολύ. Τώρα κάποια σχόλια για τις ανησυχίες ε, των ε, περιφερειών ότι θα εξασθενήσουν κάπως. Θεωρώ ξεκάθαρα ότι όταν αποφελούνται ε, ε, από χρήματα περιοχές ε, δεν θα πρέπει να υπάρχει αυτό το νότο τώρα του 2,5% αυτό δεν θα πρέπει να ισχύει για τα κράτη-μέλη που συμμετέχουν στο Συνδέοντα στην Ευρώπη. Θα πρέπει επίσης να υπάρχει δίκαιη μεταχείριση των κρατών μελών να μην υπάρχουν διαφορετικοί όροι ανταγωνισμού για αυτά τα έργα. Γι' αυτό προτείνω μια ε, διαδικασία με πολλές βαθμίδες, να γίνονται πολλές ε, προσκλήσεις και στη μέση της περίοδου να γίνεται μια αναθεώρηση όπου θα ε, αξιολογείται αν υπάρχει διακριτική μεταχείριση για κάποιες περιοχές, αν δηλαδή κάποιες περιοχές δεν παίρνουν όσα βοήθεια χρειάζεται και έτσι να μπορέσουμε να βοηθήσουμε κάποια κράτη-μέλη που επωφελούνται από τη χρηματοδότηση, ε, ώστε στο τέλος αυτά τα δέκα δις να δοθούν σωστά, ορθά, δίκαια και με ίση κατανομή και να μην επωφελείται κάποιος περισσότερο από άλλον, αλλά να υπάρχουν ίσοι όροι πρόσβασης. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά θέματα που ήθελα να θίξω. Να πω πραγματικά ότι με υπέρ αυτού του χρηματοδοτικού μέσου. Θα ήταν ε, κρίμα να πούμε ότι δεν το θέλουμε σε αυτή την Επιτροπή. Γιατί έτσι μπορεί και να χάναμε τελείως το 10 Αυτό είναι διαπραγματευτικό χαρτί για μας με το Συμβούλιο. Θέλουμε αυτά τα χρήματα, γιατί ε, οι επενδύσεις που γίνονται στα κράτη-μέλη ε, στις περιφέρειες γίνονται και αυτές επωφελούνται από τα χρήματα. Τώρα για τις ε, συνοριακές περιοχές έχουν γίνει πολλές μελέτες που βλέπουμε ότι κάθε φορά που μιλάμε για χρηματοδότηση στα διευρωπαϊκά δίκτυα, στα μέσα της Πολωνίας, στα μέσα της Γαλλίας, στα μέσα της ε, Γερμανίας εφαρμόζονται ε, έργα, αλλά αν δείτε όλο τον κατάλογο, πάλι τα ίδια θα δείτε. Δεν υπάρχει τίποτα στις διασυνοριακές περιοχές. Προτείνω λοιπόν να γίνουμε συνήγοροι στο Κοινοβούλιο των παραμεθόριων περιοχών και στην ουσία να γίνει έτσι το πράγμα ώστε πρώτα να πρέπει να πηγαίνει σε μια παραμεθόρια περιοχή ένα κόμμα της χρηματοδότησης και μετά να χρηματοδοτούνται άλλες περιοχές της χώρας. Αυτή είναι μια πολύ απτή ιδέα που ε, εξασφαλίζει ε, ακόμα λίγη δικαιοσύνη. Αυτό το μέσο λοιπόν πρέπει να το συζητήσουμε με κριτικό πνεύμα, αλλά να σκεφτούμε ότι και τελικά ίσως δεν θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε όλα τα χρήματα. Αυτό ε, συμβαίνει και με το ΕΤΠΑ. Καλό θα ήταν λοιπόν να γίνει ανακύκλωση αυτών των χρημάτων, έτσι ώστε κάποια κράτη-μέλη που θέλουν αυτά τα χρήματα για υπερπεριφερειακές ε, ε μεταφορικές διασυνδέσεις να μπορέσουν να πάνε μέσα από τα πλαίσια του, της διευκόλυνσης της συνδέοντας την Ευρώπη στα χέρια τους και έτσι νομίζω ότι θα πετύχουμε το στόχο μας. Είναι λοιπόν ένα κρίσιμο αυτό το θέμα, ένα πολύ καλό ε, ζήτημα. Ελπίζω ότι θα έχω τη βοήθειά σας και στο τέλος θα βρούμε και έναν καλό συμβιβασμό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ να περάσουμε γρήγορα στους κοιόδες. Παρακαλώ να είστε όσο γίνεται πιο σύντομα. Πιο σύντομη. Ο Βίκτορ Μποστινάρο πρώτα. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Και πάλι νομίζω ότι θα ξέρετε τι θα πω. Γιατί όλα αυτά σχετίζονται πολύ με τη δική μου έκθεση περί συνοχής και είναι και σύμφωνα με τις συζητήσεις, ε, αντιπαραθέσεις και συνεργασία που είχαμε ήδη σε αυτή την Επιτροπή. Καταρχήν να ευχαριστήσω τον κύριο Πίπερ για το τα έγγραφα εργασία του και νομίζω πως δεν υπάρχει κάποια βασική διαφωνία ή κενό ανάμεσα στη δική μου και στη δική του προσέγγιση. Πρέπει να δούμε το έγγραφο σε μια τελική εκδοχή στο τελικό κείμενο και μετά να αντιδράσουμε για το κείμενο γιατί πολλές φορές τα προβλήματα είναι στις λεπτομέρειες. Και τώρα, δεν είμαι ενθουσιώδης ε, υποστηριχτής ε, του ΣΥΕΦ για προφανείς λόγους. Όταν λοιπόν θέλουμε να επιτρέψουμε να μεταφερθούν 10 εκατομμύρια στο ΣΥΕΦ χρειάζεται δύο μεγάλες εγγύησεις. Πρώτον, τα χρήματα να χρησιμοποιηθούν για την ε, πολιτική συνοχής και όχι μόνο από την άποψη των μεταφορών, δηλαδή κοινή προσέγγιση DG Move και DG Regio. Δεύτερον, θα ήθελα εγγυήσει, σοβαρές εγγυήσει από τα κράτη-μέλη και τις περιφέρειες. Καλωσορίζω την συνοχή αλλά δεν είναι διαγωνισμός ε, ομορφιάς, ούτε διαγωνισμός ανάμεσα στις περιφέρειες και τα κράτη. Η συνοχή είναι κάτι διαφορετικό κατά τη γνώμη μου. Πρότεινα, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, και στο Γενικό Κανονισμό και στον Κανονισμό περί συνοχής θα ήθελα να προτείνω μια συμβαστική λύση που δεν είναι τέλεια, αλλά επειδή θέλω το, το να εφαρμοστεί το Ταμείο Συνοχής, γιατί συμμερίζομαι την ίδια γνώμη με τον κύριο Πίπερ, ότι μπορεί να είναι πολύ ωφέλιμο ο μέσο ώστε η Ευρώπη να αντιμετωπίσει προβλήματα που σχετίζονται με τη διασυνοριακή διάσταση. Θέλω να το δω λοιπόν να λειτουργεί και να ε, αποκομίσουμε και τα σχετικά ωφέλη. Αλλά αυτό να γίνει με πλήρε εγγυήσει. Και επίση τα κράτη-μέλη που τελικά θα είναι οι δικαιούχοι να μπορούν να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν τα προγράμματα. Γι' αυτό και προτείνω αυτή τη μεταβατική τριετή περίοδο και ζητώ από την DigiMove μείνετε ε, επίκαιροι. Θέλω ένα, ένα εφικτό, ρεαλιστικό πρόγραμμα ώστε να βοηθούν τα κρατημέλη να βοηθήσουν τις ε, διοικητικές τους και ε, θεσμικές δυνατότητες γιατί διαφορετικά ορισμένα κράτη-μέλη δεν θα μπορέσουν να εφαρμόσουν το CF και δεν θα υπάρξει ανταγωνισμός. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και αυτό είναι και το τελικό μου σχόλιο κύριε Πίπερ, όπως ξέρετε, στο Συμβούλιο γίνεται σοβαρή συζήτηση 15 κράτη-μέλη λοιπόν επισήμως δήλωσαν ότι δεν είναι ευχαριστημένοι με, με το υπάρχουν σχέδιο. Άρα λοιπόν πρέπει να δουλέψουμε για μια συμβιβαστική λύση. Εγώ θέλω να κάνω έκκληση σε όλους, DG Move, DG Regio και στους ε, συναδέλφους να δουλέψουμε για μια συμβιβαστική που θα δώσει εγγύηση αρκετή ευελιξία, θα βελτιώσει την ε, θεσμική μας, ε, τις θεσμικές μας δυνατότητες προς όφελος των περιφερειών και των κρατών μελών. Για όλους και όχι για λίγους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και να κλείσουμε τον κατάλογο. Έχουμε 7 ομιλητές, 2,5 λεπτά έκαστος. Η κυρία Μανέσκου δεν είναι εδώ. Η κυρία Κάριμα Ντέλη. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Πίπερ, σας ευχαριστούμε για την ε, παρουσίαση που κάνατε. Εγώ θα ήθελα να επανέλθω για πολλά στοιχεία τα οποία θεωρώ πολύ σημαντικά. Καταρχήν, εμείς είμαστε αντίθετοι με τα 10 δις ευρώ στο Ταμείο Συνοχής για να χρηματοδοτηθούν ε, σχέδια υποδομών μεταφορών γιατί όπως το αποδέχεται και η Κομισιόν, τα εθνικά κονδύλια δεν θα μπορέσουν να απορροφηθούν για δύο λόγους, γιατί αν δούμε από κοντά με την αρχή του use it or lose it, ή χρησιμοποίησε το ή χάσε το, η Κομισιόν μπορεί να επανεπενδύσει τα χρήματα του Ταμείου Συνοχής σε άλλα προγράμματα που βρίσκονται σε άλλα κρατημέλη που επίσης είναι επιλέξιμα για τα ταμεία συνοχής. Αυτό είναι ο πρώτος λόγος. Η Κομισιόν βεβαιώνει πως κανένα επιλέξιμο κράτος μέλος για το Ταμείο Συνοχής ε, δεν θα μείνει χωρίς ε, σχέδιο. αυτό δεν σημαίνει πως τα κονδύλια ε, του Ταμείου θα χρησιμοποιηθούν ισότιμα. Άρα λοιπόν η Κομισιόν εδώ ακολουθεί περισσότερο τη λογική του αριθμού των σχεδίων και όχι τα ποσά των ποσών Επιπλέον, η προσαρμογή της Κομισιόν για να λάβει υπόψη όσο γίνεται περισσότερο τα, τα εθνικά κονδύλια για τα ταμεία συνοχής, έτσι ώστε κανένα κράτος μέλος να μην ε, τιμωρηθεί. Και αν σκεφτούμε ότι ε, ψηλά ποσοστά σε χρηματοδότηση είναι απαραίτητα στις χώρες, θεωρώ ότι το να πάρουμε αυτά τα χρήματα στο Ταμείο Συνοχής είναι ε, σφάλμα, γιατί ένα κράτος μέλος το οποίο θα αφιερωνό, θα έβλεπε το δικό του κομμάτι του συνοχής να αφιερώνεται σε ένα άλλο κράτος μέλος, ε, θα δει ότι τα χρήματά του θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε άλλα προγράμματα συνοχής στη δική του επικράτεια. Ευχαριστώ πολύ κυρία Ντέλη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εξ ονόματος της επιτρέψτε μου να πω δύο-τρία πράγματα. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον κύριο Πίπερ, τον εισηγητή. Η ομάδα μας έχει πει πολλές φορές και θα επιμείνουμε ότι δεν είμαστε κατά της δημιουργίας ενός νέου μέσου, αλλά πιστεύουμε ότι χρειαζόμαστε μία πολιτική που θα είναι σε θέση να υποστηρίξει σε θέματα ενέργειας και μεταφορών, μεταξύ άλλων, διευρωπαϊκά. Ε, πιστεύουμε όμως ότι για να μπορέσουμε να το επιτύχουμε αυτό, αυτά τα δέκα συμπληρωματικά δις από το Ταμείο Συνοχής λανθασμένα θα χρησιμοποιηθούν εδώ. Πιστεύουμε ότι έτσι κατά κάποιο τρόπο πετάμε 26. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν με την Κομίσιο κατά πόσον θα μπορέσουμε τον το Επίσης, η γραμματεία είναι αυτή η οποία θα πάρει την τελική απόφαση και τα κράτη-μέλη δεν θα έχουν σχεδόν καθόλου δυνατότητα επηρεασμού αυτής της απόφασης. Όπως είπε και ο κύριος Όλμπρεχτ, η δημιουργία αυτό το Connecting Europe, συνδέοντας την Ευρώπη του προγράμματος, καλή φαίνεται, αλλά το ερώτημα είναι πώς σχεδιάζει να κάνει κάτι τέτοιο η Κομισιό με τα κονδύλια αυτά που θα πάρει από τα μη Θα θέλαμε να έχουμε λεπτομέρειες για το πώς θα ενεργήσει. Θα ήθελα να ζητήσω από τον κύριο Πίπερ, τον εισηγητή, να λάβει υπόψη την επιλεξιμότητα του ΦΠΑ και το κόστος αυτό το οποίο είναι σημαντικό είναι οι σιδηροδρομικές ε, συγκοινωνίες που είναι πάρα πολύ σημαντικές για τις νέες χώρες. Θα σας είμαστε ευγνώμονες αν το λαμβάνατε αυτό υπόψη κύριε εισηγητά. Και ελπίζουμε ότι κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων θα μπορούσαμε να ζητήσουμε από τον εισηγητή να είναι ε, μαζί μας. Αντικαθιστά κανείς τον Τζον Μπάφτον ή την Κορνέλια, όχι. Τον Γιώκιμ Τσέλλαρ το δίνω μέσα στο λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς ευχαριστώ Μάρκους για το έγγραφο εργασίας ε, που ε, έχει πολύ συγκεκριμένη δουλειά γίνει ε, σε σχέση με αυτή, αυτό το εργαλείο. Πρόκειται για μια νέα αρχή που θα πρέπει να έχει 50 δις ευρώ. Μια νέα αρχή η οποία θα πρέπει να υπόκειται στην Επιτροπή του Προϋπολογισμού και τα 10 ε, δις ε, θα πρέπει να πάνε στις χώρες συνοχής μέσα από το Ταμείο Συνοχής. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Γιατί αυτή η διευκόλυνση συνδέοντας στην Ευρώπη δημιουργήθηκε γιατί για δεκαετίες, για χρόνια μιλάμε και συζητάμε για ευρωπαϊκά διασυνοριακά δίκτυα τα οποία τελικά δεν πραγματοποιούμε. Και υπάρχουν τώρα τρεις προτεραιότητες. Ε, τηλεπικοινωνίες, ενέργεια, υποδομή και μεταφορές, ε, συνδρομικές κτλ. Ε, και δημιουργία των αντίστοιχων διαδρόμων ο τρόπος εργασίας αυτού του ε, μέσου για μένα είναι περί... σκοτεινός. Στις ε, τηλεπικοινωνίες έχουμε μεγάλες ιδιωτικές ε, εταιρείες. Τα κίνητρα εδώ όμως θα πρέπει να δοθούν από τα κράτη σε αυτή τη διευκόλυνση. Και πώς θα λειτουργήσει αυτό με ξεπερνά. Ε, πάντως 10 ε, δις προβλέπονται στη Γερμανία μόνο για την ενεργειακή υποδομή και τα αντίστοιχα δίκτυα ηλεκτροδότησης. Μιλάμε για 130 δις ευρώ που χρειάζονται. Φαντάζεστε τώρα σε σχέση με τα 10 δις τι διαφορά υπάρχει και άλλα 300 και άλλα 30 για την υποδομή μεταφορών. Αυτό έχει να κάνει με δίκτυα ε, και με σιδηροδρομικές γραμμές σε μικρές περιοχές της Ευρώπης και γι' αυτό θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ε, εάν θα είναι αυτοί που λειτουργούν τις υποδομές αν ε, αυτοί που λειτουργούν τις υποδομές και οι επενδύσεις που κάνουν ε, τα κράτη-μέλη ε, συμφωνούν με το πλαίσιο. Και σε επίπεδο σχεδιασμού θα πρέπει να μιλήσουμε και γι' αυτό, αν υπάρχει τέτοιο σχεδιασμός δηλαδή στις περιφέρειες ε, και στα κράτη, γιατί αυτό θα αποτελούσε πρόβλημα στην πραγματοποίηση αυτού της πολύ καλής λύσης που έχει δημιουργηθεί με πολύ καλές προθέσεις, αλλά το αν θα πραγματοποιηθεί τελικά δεν, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Ε, νομίζω ότι τα δέκα δις ε, για τις χώρες συνοχής ε, θα πρέπει να αποφασίσουν οι χώρες αυτές αν τα θέλουν ή όχι για τη διευκόλυνση ή όχι. Τέλος πάντων είναι μια πραγματικότητα, μια συζήτηση. Συμφωνώ με τον Γιάνν Όλμπριχτ. Καταρχάς δεν συνδέεται άμεσα με τον κανονισμό για τα ε, διαρθρωτικά ταμεία αυτή η διευκόλυνση. Η μόνη σχέση με αυτόν είναι τα 10 δις για το Ταμείο Συνοχής. Και αν η Κομισιόν και το Συμβούλιο και τα κράτη-μέλη συμφωνήσουν για τη βάση αυτής της αρχής με αυτά τα χρήματα μέχρι το 2020 ε, και αν θέλουν να, να τα καταφέρουν βέβαια. Αν δεν μπορούν, παρακαλώ πρέπει να τα εξετάσουμε και πάλι και τελικά να, ε, το, να εντάξουμε αυτό τη διευκόλυνση στο πολιετές ε, δημοσιονομικό πλαίσιο. Ευχαριστούμε τον Γιώχημ. Ε, dziękuję bardzo. Ε, chcę podziękować również sprawozdawcy za ε, przedstawiony dokument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 καθώς και την κατανομή του κεφαλαίου στα πλαίσια των PPPs, των εταιρικών σχέσεων ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, Και αυτά δεν θα πρέπει να είναι επωφελή για τους πολίτες. Τώρα, ίσως είναι λυπηρότητα δέκα δις. Θα φύγουν από το Ταμείο Συνοχής από τη μια. Αλλά από την άλλη υπάρχουν περιοχές που είναι πανευτυχείς που θα διατεθούν κάποια από αυτά σε αυτές και θα τα χρησιμοποιήσουν σε άλλους τομείς μεταφορά ενέργειας, ε, μεταφορές λοιπά. Όπου εδώ χρειάζονται έργα βελτίωση. Ευχαριστώ. Οι δύο συνάδελφοι από την ε, Επιτροπή, ο κύριος Πακέ είναι εδώ. Ποιος θέλει να μιλήσει πρώτος. Ο πρώτος ο κύριος Πακέ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολύ σύντομα για να ευχαριστήσω για την έκθεσή τον κύριο Πίπερ που αντικατοπτρίζει σωστά τον στόχο της πρότασης Επιτροπής που όντως είναι να είναι συμπληρωματικό το Connecting Europe Facility με τα υπάρχοντα μέσα τα και τα προτινόμενα μέσα στα πλαίσια της περιφερειακής ανάπτυξης και της συνοχής. Άρα το Connecting Europe είναι οριζόντια εφαρμόσιμη και των, μεταξύ των διαφόρων υπηρεσιών η COM και η MOVE και η REGIO είναι υπεύθυνε και αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να εξασφαλίσουμε ότι η συμπληρωματικότητα των δύο αυτών προγραμμάτων θα οδηγήσει σε μεγάλες συνέργειες. Δεν θα μπω τώρα σε λεπτομέρειες, διότι τις γνωρίζετε. Η Επιτροπή δαπάνησε σε ανώτερο επίπεδο μεγάλη πόσα ενέργειας για να συζητήσει με τα κράτη-μέλη, για να δει πώς θα αναπτυχθούν αυτά τα σχέδια, τι θα γίνει με αυτά τα δέκα δις. Και βλέπουμε από την συζήτηση ότι υπάρχει μια κάποια ανησυχία που εκφράζεται σε πολιτικό επίπεδο, αλλά νομίζω ότι όλη η τεχνική δουλειά που έγινε μπορεί να αποδείξει κυρίως τους υπεύθυνους των μεταφορών ότι η Επιτροπή θέλει να εφαρμόσει την, ε, με απόλυτη προτεραιότητα το θέμα που αφορά εθνικά σχέδια σε θέματα μεταφορών που θα παρουσιαστούν. Χαιρετίζω τις συστάσεις του κυρίου Πάιπερ, ώστε μετά το 2014 να συνεχίσουμε με νέους μειοδοτικούς διαγωνισμούς, ώστε να μπορέσουν να προετοιμάσουν και να υποβάλουν όλα τα κρατημέλη καλά σχέδια και να καταλήξουμε σε όριμα και ποιοτικά σχέδια τα οποία θα επιλεγούν ώστε όταν τα επιλέξει η Επιτροπή να είναι σίγουροι ότι ε, θα έχουμε μεγάλη συνέργεια και συνεργασία μεταξύ των χωρών που επιλέγονται στα πλαίσια του Connecting Europe και ότι θα δοθεί προτεραιότητα σε δικά σχέδια. Για να απαντήσω στον κύριο Μποστινάρου. Ίσως θα μπορούσαμε να είμαστε και πιο ακριβείς ώστε να μπορέσουν να βοηθούν περισσότερο συνάδελφοι νέων κατών. Θα δώσουμε περισσότερες οδηγίες για να γνωρίζουν όλοι πώς θα λειτουργήσει αυτό το σχέδιο. Τώρα, όσον αφορά την οριμότητα, έχετε μια σειρά προγραμμάτων που θα πηγαίνει μαζί με το Connecting Europe, που θα πάει στο Συμβούλιο τις 7 Ιουνίου υπήρξε συμφωνία εκ μέρους των Υπουργών. Πρόκειται για κατάλογο στον οποίο προσθέθηκαν κάποια έργα. Δεν είναι ευχολόγιο, αλλά είναι προτεραιότητες των εταίρων μας τις χώρες με τις οποίες συνεργαζόμαστε και έργα τα οποία φαίνεται ότι έχουν οριμάσει και μπορούν να εφαρμοστούν. Πολλές φορές κάποια είναι στην πρώτη φάση, στην προπαρασκευαστική, άλλα έχουν οριμάσει περισσότερο Έχουμε λοιπόν ε, μία καλή βάση που θα μας επιτρέψει να προχωρήσουμε και έτσι να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα δέκα πολύ καλά σε όλες τις χώρες της συνοχής. Τώρα να αφορά το κάπινγκ που ανέφερε ο εισηγητής, είναι θέμα MFF. Δεν έχει σχέση με το Connecting Europe, αλλά είναι πολύ λογικό το επιχείρημα το οποίο υπάρχει στην έκθεση και θα ευρεθεί εκ μέρους των θετικών οργάνων μια κάποια λύση. Τώρα, όσον αφορά τις διασυνοριακές περιοχές, συμμερίζομαι την εκτίμηση που έγινε πρόκειται για co-mission, για μια κοινή αποστολή που έχουμε, δηλαδή να μπορέσουμε σε αυτό το ευρωπαϊκό δίκτυο να συνενώσουμε ε, πόλεις που βρίσκονται ε, σε όμορες περιοχές και από ό,τι γνωρίζω από την ε, ε, εμπειρία που έχουμε από το TEN-T, τα περισσότερα σχέδια βρίσκονται σε τέτοιου είδους περιοχές και θα πρέπει και πάλι να εξετάσουμε τον κατάλογο να εξασφαλίσουμε ότι όλα αυτά αντικατοπτρίζονται καλύτερα στο πρόγραμμα και στην ιδέα να χρησιμοποιήσουμε κονδύλια από το TNT και από τις διασυνοριακές περιοχές. Αυτά τα ποσά όντως είναι το ελάχιστο το οποίο θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε για τα IT και τις ε, μεταφορές και αν είχαμε περισσότερο θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε περισσότερα σχέδια σε πολλές χώρες. Ευχαριστώ. Αυτά ήθελα να πω προς το παρόν. Δεν έχω πολλά να προσθέσω, Πρόεδρε. Απλώς θα ήθελα να τονίσω ότι χρειάζεται να υπάρχει κοινή προσέγγιση. Και κατά την άποψή μας αυτό αντικατοπτρίζεται και στους κανονισμούς και στα, σε άλλα μέσα, στο CSF. Εκεί λέγεται και εξηγείται πώς θα δουλέψουν από κοινού αυτά τα ταμεία. Θα πρέπει όμως, όπου μπορούμε, να θέσουμε μέσω των εταιρικών συμφωνιών ε, σε εφαρμογή του κανονισμού, διότι εδώ το πιο σημαντικό θέμα είναι η διασύνδεση μεταξύ των πιο, κυριο... των πιο σημαντικών project όπου χρηματοδοτούνται μεγάλα έργα υποδομής και άλλα που θα χρηματοδοτούν από το Connecting Europe και τα πιο σημαντικά project θα πρέπει να συμπεριληφθούν σε έναν κατάλογο ώστε να κάνουν την επιλογή τους τα κράτη-μέλη για έργα τα οποία θα μπορέσουν να χρηματοδοτηθούν και από το Connecting Europe. Το λέγω αυτό διότι θα πρέπει να επιτύχουμε πολύ καλή συνεργασία και συντονισμό. Το Partnership Agreement, η συμφωνία Εταιρική, να φέρει και τι θα είναι θέμα προτεραιότητος και τι ETC και στα πλαίσια των προγραμμάτων ETC μπορούμε και έργα υποδομής να χρηματοδοτήσουμε και η Ισχύει εδώ η εξαίρεση των, σχεδίων mainstream. Τώρα όσον αφορά το κάπινγκ. Αυτό που πρέπει να έχουμε κατά νου είναι ότι η συλλογιστική του κάπινγκ αφορά το θέμα της απορρόφησης των κονδυλίων. στα πλαίσια του Connecting Europe. Ευχαριστώ. Ο Μάρκος Πάιπερ. Ευχαριστώ την Επιτροπή. Ο Μάρκος Πάιπερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Λίγο με εκπλήσει ότι εξ αρχής ε, χαιρετάτε αυτό το, και καλωσορίζετε αυτό το ε, εργαλείο. Μόνο μία πολιτική ομάδα είπε ότι πάει προ λάθο κατεύθυνση. Έχουμε οπότε μία καλή βάση για να συμφωνήσουμε σε ένα συμβιβασμό όπου κάποια κεντρικά σημεία δεν είναι συζητήσαμα. Ίσως θα πρέπει να ψηφίσουμε ο καθένας όπως, ε, πρέπει, όπως θέλει, ε, γιατί υπάρχει αυτό το θέμα του ανταγωνισμού, η διαδικασία του ανταγωνισμού πρέπει οπωσδήποτε να βρίσκεται εδώ και οπωσδήποτε οι παραμεθόρες περιοχές ε, είναι κάτι που εμένα με ενδιαφέρει να στηρίξω. Άρα, πέρα από αυτά, νομίζω ότι γενικά θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε γρήγορα. Ένα τελευταίο θέμα που έχει να κάνει με τον νέα αυτή αρχή, τον νέο φορέα. Σε κάθε ευκαιρία και εγώ βρίζω τους, όλους τους φορείς ε, τους ευρωπαϊκούς. Αλλά για μία πρώτη φορά εδώ έχουμε κάτι που ε, μας οδηγεί σε, μια δεσμευτική, σε ένα δεσμευτικό συντονισμό ε, μεταξύ των κρατών έτσι ώστε σε κάθε χώρο να υπάρχει μια καλή ε, αξιοποίηση των δυνατοτήτων. Για πρώτη φορά που είναι, ήρθε η στιγμή να πούμε ότι πρέπει να κάνουμε κάτι για κάποιες συγκεκριμένες περιοχές. Πραγματικά είμαι απόλυτα της άποψης ότι αυτό έχει νομιμοποίηση και πραγματικά ελπίζω ότι θα συνεννοηθούμε για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον Μάρκους. Ε, με αυτό κλείνουμε το σημείο 4 της ημερήσιας διάταξης και περνάμε στο σημείο 5 της σα διάταξης, θέσπιση προγράμματος για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα. Πατρίς Τυρόλιν, έχετε το λόγο. Ε, Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, το πρόγραμμα LIFE είναι το κύριο μέσο άμεσης χρηματοδότησης της κοινοτική πολιτικής προστασίας του περιβάλλοντος, βιοπικιλότητας και της ε, ε, προσαρμογής στις κλιματικές αλλαγές στα πλαίσια της στρατηγικής 2020. Η πρόταση αυτή της Επιτροπής περιέχει τρία κυρία στοιχεία. Ενσωματωμένα σχέδια, ΦΠΑ και ποσοστό χρηματοδότησης παρά το γεγονός ότι υπάρχει αύξηση των κονδυλίων, το πρόγραμμα LIFE υποχρηματοδοτήσει αν δούμε ποιες είναι οι απαραίτητες επενδύσεις που πρέπει να γίνουν για να υλοποιηθούν αυτοί οι στόχοι. Για το λόγο αυτό υποστηρίζω την πρόταση της Επιτροπής ότι θα πρέπει να υπάρξουν ε, ενοποιημένα και ενσωματωμένα σχέδια και να βελτιωθούν οι συνέργειες μεταξύ πολιτικής συνοχής και προγράμματων LIFE. Οι δράσεις αυτές θα είναι εποφελής από την Προγραμματομοσύνη την οποία έχει ήδη η Επιτροπή Περιβάλλοντος και από τα κονδύλια των Ταμείων Συνεχής. Πιστεύω παρόλα αυτά ότι θα πρέπει να κάνω τις εξής παρατηρήσεις. Θα πρέπει να είναι αποδοτικές οι συνέργειες και θα πρέπει να υπάρξουν μηχανισμοί συντονισμού μεταξύ των διαφόρων μετεχόντων στα θέματα αυτά. Παρά το γεγονός ότι το πρόγραμμα LIFE πρέπει να ανταμείψει σχέδια ε, τα οποία έχουν αναπτυχθεί τοπικά, θα πρέπει να μπορέσουν τα προγράμματα που θα επωφεληθούν εδώ να είναι γεωγραφικά ισορροπημένα, ώστε όλα τα κράτη-μέλη να υποφεληθούν πλήρως. Εξάλλου, είμαι κατά της, ε, ε, το αποκλεισμού της ΦΠΑ και των δαπανών για το προσωπικό που θα ασχοληθεί με το live, δεδομένου ότι οι επιπτώσεις ενός τέτοιου μέτρου φαίνεται ότι τελικά με αυτά τα στοιχεία θα αποβεί αρνητικό. Επίσης, νομίζω ότι είναι πρωταρχή σημασία στα πλαίσια του ΙΝΑΤΟΥ να διατηρήσουμε κάποιες βασικές αρχές δημοσιονομικών κανόνων, όπως αυτούς που ακολουθούμε στα πλαίσια της πολιτικής συνοχής. Κατά συνέπεια, θα ήθελα να επανέλθουμε στα προηγούμενα ποσοστά συγχρηματοδότησης για να εγγυηθούμε στην δημοσιονομική ισορροπία ε, συνέχεια. Εξάλλου, ποστίβω ότι είναι πολύ σημαντικό να έχουμε μία ε, προσέγγιση η οποία θα μπορέσει να ωφελήσει την ενότητα των σχεδίων σε όλες τις χώρες. Επίσης θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με σχέδια τα οποία θα παρουσιάσουν ε, τα πιο απομεξιμένες ε, περιοχές της Ευρώπης. Θα πρέπει να επενθυμίσουμε επίσης στην Γενική Διάθεση Περιβάλλοντος να τιμήσει τις υποχρεώσεις της. Πιστεύω θα ήταν σκόπιμο επίσης να αυξήσουμε τα ποσοστά συγχρηματοδότης για κάποιες προβληματικές περιοχές που έχουν ευαίσθητα ή οικοσυστήματα για ορεινές νησιώτικες περιοχές που έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και επηρεάζονται ιδιαίτερως από τις κλιματικές αλλαγές. Συμπερασματικά θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα μέλη της γραμματείας μας, καθώς και τους ε, ε, βοηθούς που που με βοήθησαν να κάνω την έκθεσή μου και περιμένω τις παρατηρήσεις των συναδέλφων. Δεν βλέπω κανένα από τους σκιώδεις ηγητές. Ίσως εδώ, αν δεν υπάρχει κανείς, ο κύριος Σομαλζή να πάρει το λόγο παρακαλώ. Madame Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να χαιρετήσω την ε, ποιοτική εργασία του συνάδελφου Πατρίστη Ρολιά. Κυρίως θα ήθελα να ευαισθητοποιήσω τους συναδέλφους της Επιτροπής Ρέτζι σε ένα θέμα. Οι πάρα πολύ απομακρυσμένες περιφερειακές γαλλικές περιφέρειες της Γαλλίας αποκλείονται από το Natura 2000 και κατά την άποψή μου θα πρέπει να διαρωτηθούμε πρόβλημα υπάρχει. Το πρόβλημα το οποίο ανέφερα στην Επιτροπή, υποβάλλοντας γραπτή ερώτηση που είναι στη διάθεσή σας. Και μου απήντησε βέβαια η Επιτροπή. Περί τίνος πρόκειται. Η πανίδα, η χλωρίδα, οι βιότοποι των δικών μας περιοχών δεν συμπεριλαμβάνονται στην ε, οδηγία Natura 2000. Άρα εξορισμού αποκλειόμεθα από κάποια προγράμματα που προβλέπει το LIFE και το Natura. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να ασχοληθούμε με αυτό το θέμα. Γιατί δεν βλέπω για ποιο λόγο στις περιοχές μας, στις οποίες υπάρχει μεγάλη βιοπικιλότητα και τα κυριότερα είδη, χλωρίδα, πανίδα, πτηνά και ό,τι θέλετε, να μην τα συμπεριλαμβάνουμε στο Natura 2000. Βεβαίως, είμαι υπέρ της πρότασης για το live που κάνει ο εισηγητής, ώστε τα TomDom να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα αυτό. Εγώ κατέθεσα κάποιες τροπολογίες, ώστε να συμπεριληφθεί εδώ το μήνυμα του νησιού της Ρεϊνιό. Δηλαδή το μήνυμα που είχε, η δήλωση δηλαδή που είχε παρουσιαστεί μετά από την διάσκεψη που έγινε κατά τη διάρκεια της Γαλλικής Προεδρίας Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Ρεϊνιό. Δεδομένου ότι εδώ έχουμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα βάση εργασίας και η δυνατότητα να προχωρήσουμε στη συγκεκριμενοποίηση των ε, προτάσεων που είχαν γίνει τότε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Λόι. Σας ευχαριστώ πολύ. Η σκιώδης μας δεν είναι εδώ, οπότε απλώς θα σας παραθέσω τις ε, παρατηρήσεις της. Καταρχήν να ευχαριστήσω τον κύριο Τυρολιά που προχώρησε το θέμα όσον αφορά την περιφερειακή διάσταση Εξάλλου, ο δεύτερο στόχο των όσων κάνουμε στην Ευρώπη 2020 είναι να προχωρήσουν ακριβώ αυτά τα μέσα στον περιφερειακό σχεδιασμό. Βάση περιπτώσει, πρόκειται για χωριστό πρόγραμμα. Επίσης υπάρχουν ένα-δύο παρατηρήσεις που κάνουμε ότι καταρχήν θα δείτε το ίδιο με τις ε, κατεξιδότητες συμπράξεις και το θέμα είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει σωστή ισορροπία ανάμεσα στο τι περιλαμβάνεται στο νομικό κείμενο και στο τι θα κάνει μετά η ε, κομισιόν. Για την επιλεξιμότητα και τους δημοσιονομικούς κανόνες είναι σημαντικό να ακολουθούνται οι ίδιες μέθοδοι και οι ίδιες σχέσεις ανάμεσα στους δικαιούχους και τον επίσημο σχεδιασμό και τις αρχές πληρωμών. Έτσι, Θα έχουμε όσο γίνεται περισσότερα στοιχεία όσον αφορά την επιλεξιμότητα και τους κανόνες. Αυτό που κάναμε σε σχέση με την πρόταση είναι η προσέγγιση της επικουρικότητας. Να έχουμε δηλαδή πλήρη συνεργασία σε σχέση με τα όσα κάνουμε ώστε να έχουμε μια πιο πράσινη και βιώσιμη προσέγγιση στην περιφερειακή πολιτική. Έτσι να δώσουμε μια θετική εικόνα. Δεν βλέπω κάποιον άλλον να θέλει να πάρει το λόγο, οπότε θα ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν θέλουν να σχολιάσουν. Ο κύριος Μαχτά. Σας ευχαριστώ. Καλησπέρα σε όλους. Θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας ε, τους εισηγητές ε, για την ε, χρήσιμη συμβολή τους στη συζήτηση. Θα ήθελα να θυμίσω στους ευρωβουλευτές ότι η Κομισιόν προτείνοντας αυτό το νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης πολιτικών του περιβάλλοντος και καταπολέμησης των κλιματικών αλλαγών θέλησε να προσεγγίσει το τρέχον πρόγραμμα με την εφαρμογή των πολιτικών και να το χρησιμοποιήσει για να διευκολύνει ε, για την ένταξη των ε, πολιτικών περιβάλλοντος στις υπόλοιπες πολιτικές της Ένωσης. Γι' αυτό και θέλω να χαιρετήσω τις βασικές γραμμές της έκθεσης του κυρίου Τυρολιά. Ωστόσο, αν μου το επιτρέπετε κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να κάνω κάποιες σύντομες παρατηρήσεις το πρώτο που θα ήθελα να πω είναι ότι ευχαριστώ τον εισηγητή για τη στήριξη για τα ολοκληρωμένα προγράμματα που στην ουσία επισημοποιεί την επιθυμία της Κομισιόν για να έχουμε τα απαραίτητα εργαλεία στο πλαίσιο του προγράμματος για τη διευκόλυνση τη ένταξη των περιβαλλοντικών θεμάτων στι υπόλοιπε πολιτικέ και γι' αυτό και ευχαριστώ την Επιτροπή Ρέτζη για τη στήριξή του στην ευθυγράμμιση και την εφαρμογή της πρότασης και των διατάξεων μέσα στο πλαίσιο του γενικού, κοινού μάλλον στρατηγικού προγράμματος, πλαισίου, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η συνοχή αυτού του προγράμματος με τα υπόλοιπα στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για τις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές. Επιπλέον πρέπει να κάνουμε και κάποιες παρατηρήσεις σε σχέση με τις προτάσεις που έγιναν από τον εισηγητή ε, όσον αφορά τη διεύρυνση των τομέων που θέλει ο εισηγητής για τα ολοκληρωμένα προγράμματα σε τομείς όπως η ποιότητα του ε, θαλάσσιου νερού ή η ποιότητα των εδαφών. Ξέρω ότι δεν έχουν συζητηθεί οι προπολογισμοί και δεν έχουν ακόμα οριστικοποιηθεί. Ε, Κάνα την παρατήρηση αυτή και στην Επιτροπή της Περιβάλλοντος σήμερα το πρωί, αλλά το να θέλουμε να διευρύνουμε τους ολοκληρωμένα προγράμματα σε άλλους τομείς δεν σημαίνει ότι απαραίτητα θα συνοδευτεί και από αυξημένα κονδύλια. Θα θέλαμε βέβαια και η Κομισιόν θα το ήθελε, αλλά θα πρέπει να ξέρουμε ότι για τα ολοκληρωμένα προγράμματα η Κομισιόν σε χρηματοδότηση σχετικά ψηλή για να μπορέσει να διευκολύνει όντω αυτό το εφέ μόχλευσης. Επιπλέον, όσον αφορά την εφαρμογή του προγράμματο, το LIFE γνωρίζει επιτυχία εδώ και 20 χρόνια, το διαχειρίζεται κεντρικά η Κομισιόν. Υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση από ό,τι δυνατότητε, ε, δυστυχώ, και μάλιστα η ζήτηση αυξάνεται τα τελευταία χρόνια. Η επιθυμία του εισηγητή να έχει ποσοστό συγχρηματοδότηση ειδικό για κάποιε ζώνε διοπικιλότητας ή λιγότερο προνομιού και ζώνες όσον αφορά το οικονομικό επίπεδο που κατανοούμε βέβαια την αρχή αλλά τίθεται το θέμα της εφαρμογής γιατί η λιγοτερο προνομιουχε ε, ζωνες οσον αφορα το οικονομικο επιπεδο που κατανοουμε με βεβαια την αρχη αλλα τιθεται το θεμα της εφαρμογη γιατι η κομισιον χειριζεται με τον ίδιο τρόπο και ισότιμο τρόπο όλα τα προγράμματα live και είναι δύσκολο να τροποποιηθεί το ποσοστό συγχρηματοδότησης για συγκεκριμένα προγράμματα γιατί δεν μπορούσαμε να παρακολουθήσουμε γιατί εν γέννη πρόκειται για τις υπερπεριφερειακές, τις ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιφέρειες δηλαδή ε, και έπειτα για τις μη προνομιούχες και τις προνομιούχες περιοχές ποιος θα ήταν το ποσοστό συγχρηματοδότησης υπάρχουν θέματα σκοπιμότητας δηλαδή και σε αυτά θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας τώρα. Τα γνωστά εδάφη και της Γαλλίας, τα υπερπόντια, και εκεί θελήσαμε να μπορέσουν να γίνουν πολιτικές εφαρμογής διαπραγμάτευσης και μεταγραφής των, περιβαλλοντικών πολιτικών και εκεί σε εδαφικό επίπεδο και αυτό υπογραμμίστηκε από ε, τους ε, κύριους βουλευτές, όλα τα κράτη και όλες οι περιφέρειες δεν είναι στο ίδιο επίπεδο όσον αφορά την μεταγραφή και την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου, γιατί εκεί γίνεται διάκριση ανάμεσα σε δύο περιφέρειες, τις ε, ιδιαίτερα απομακρυσμένες και τα υπερπτώντια εδάφη, όπου η νομοθεσία διαφέρει. Ας πούμε, για το Natura 2000 η οι υπερπεριφερειακές ε, περιφέρειες ε, φαίνεται να αποκλείονται. Όμως, επειδή χαίρουν του κοινοτικού δικαίου, χαίρουν των προγραμμάτων LIFE. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο η Κομισιόν σκέφτεται εναλλακτικέ λύσεις φυσικά. Ακριβώς έτσι ώστε να υπάρχει αυτή η ιδιαίτερη μεταχείριση για αυτές τις ε, περιφέρειες και εδάφη, τα υπερπόντια Προσπαθούμε να βρούμε το πιο σωστό τρόπο ώστε να μπορέσουν να ωφεληθούν αυτές οι περιφέρειες από οικονομική στήριξη, αλλά σίγουρα όχι στο πλαίσιο του LIFE, ίσως ε, από το Ταμείο Ανάπτυξης ή κάποια άλλη επιλογή. Ακόμα το σκέφτεται η Κομισιόν. Νομίζω ότι κάλυψα τις παρατηρήσεις και μπαίνω στη διάθεσή σας αν υπάρχουν ερωτήσεις. Κύριε Τυρολιά, θέλετε να απαντήσετε ή να σχολιάσετε για να κλείσουμε το θέμα. Όχι, άκουσα τα διάφορε διάφορες ε, που εκφράστηκαν για τη διάρκεια αυτή της συζήτηση. Οι απαντήσει ήταν ικανοποιητικέ. Υπάρχουν βέβαια και κάποιοι τομεί που θα πρέπει ίσως να τολμήσουμε να κάνουμε κάτι παραπάνω. Αλλά θα ήθελα να λάβω υπόψη όλες τις ε, παρατηρήσεις που έγιναν και αναμένω και προτάσεις ε, τροπολογιών από τους συναδέλφους και είμαι σίγουρη ότι θα βρούμε μια γενική συνένεση για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Η μόνη υπόφαση που πρέπει να λάβουμε τώρα είναι να αποφασίσουμε για την προθεσμία υποβολή τροπολογιών που θα είναι σύντομη λόγω τη ψηφοφορία που θα γίνει στην Επιτροπή Περιβάλλοντος πριν από την συνάντησή μα το Σεπτέμβριο. Άρα πρέπει να ψηφίσουμε τον Ιούλιο, γι' αυτό και η προθεσμία υποβολή τροπολογιών είναι η 22 η Ιουνίου στις 12 μεθαύριο. Και τώρα θα ήθελα να περάσουμε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης, το κυρίας Βέσφαλ, που είναι η Ευρωπαϊκή Στατιστική και η Δημογραφία. Εξέταση του σχεδίου γνωμοδότησης. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Δεν ε, είμαι ειδική στην δημογραφία, και στα δημογραφικά δεδομένα, αλλά είναι καλό που μπόρεσα να κάνω αυτή την έκθεση μαζί με τους κοιότητες ηγητής. Έχει να κάνει ε, με την ε, εναρμόνιση των δεδομένων ε, για τον πληθυσμό. Πρόκειται για ένα πλαίσιο για συστηματική έκδοση στατιστικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη δημογραφικά, με δημογραφική διάσταση στατιστικά στοιχεία για τον πληθυσμό, για τις γεννήσεις, τους θανάτους κτλ. Ε, καλωσορίζω την ε, θέληση για εναρμόνιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και την χρήση στατιστικών στοιχείων για το θέμα ε, ε δημογραφικών στατιστικών. Ε, αυτό παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο με τα στατιστικά στοιχεία μπορούμε να καταφέρουμε να κάνουμε συγκρίσεις ε, και να βγάλουμε συμπεράσματα τα οποία είναι σημαντικά ε, γιατί μας ανοίγουν ε, διάφορους δρόμους και επιλογές. Δεν χρειάζεται να σας θυμίσω ότι τα τελευταία χρόνια υπήρχε μια έκθεση πρωτοβουλίας για τις δημογραφικές αλλαγές που ψηφίστηκε με γνώμονα και τη μελλοντική υποτιλητική συνοχής. Έτσι λοιπόν έχουμε πάντοτε αναφερθεί στη σημασία αυτού του θέματος των στατιστικών. Με αυτή την έκθεση απαιτείται οι δημογραφικές αλλαγές στις διάφορες περιφέρειες να αντικατοπτρίζονται στις στατιστικές. Έχουμε τοπικές, ε, περιφερειακές και εθνικές βάσεις δεδομένων ε, για τις δημογραφικές αλλαγές που θα πρέπει να είναι συγκρίσιμες έτσι ώστε να μπορούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο να αξιολογούνται τα στοιχεία και να γίνεται ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των ε, περιφερειών και των δήμων, ας πούμε. Όταν κάτι τέτοιο μπορεί να εφαρμοστεί, πρέπει να εφαρμοστεί σε τεχνικό επίπεδο, ε, θα χρειαστεί ε, περαιτέρω υποστήριξη. Αγαπητοί συνάδελφοι, να μιλήσω για ένα ακόμα θέμα σύντομα. Στην πρόταση θέλει η Κομισιόν ε, να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία για την δημιουργία δικτών. Αυτό το υποστηρίζω περίφραστα. Ο δείκτης δημογραφικής ευπάθειας μπορεί να είναι ένας δείκτης αυτού του είδους ε, στην ε, ε, έκθεση. Ακριβώς αυτό απαιτούμε, να χρησιμοποιείται τακτικά αυτός ο δείκτης και αυτό να είναι αναγνωρίσιμο. Δηλαδή ποιες είναι οι περιφέρειες της Ευρώπης που έχουν μεγάλες δημογραφικές αλλαγές. Επίσης υποστηρίζω γι' αυτό το λόγο την πρόταση της Κομισιόν στην πρώτη ε, ε, γραμμή αναφέρονται οι κανόνες εφαρμογής. Ε, η ανησυχία ότι για κάποιες περιφέρειες μπορεί να υπάρχει πάρα πολλή δουλειά που θα πρέπει να γίνει με τη συλλογή των στοιχείων. Τώρα δεν ισχύει γιατί το άρθρο 3.1 επιτρέπει στενότερη προσέγγιση. Οι τροπολογίες μου για την ε, Επιτροπή Περιφερειών έχουν να κάνουν ακριβώς ε, με το ρόλο των περιφερειών σε αυτή τη διαδικασία. Να περιλαμβάνονται στις ε, στατιστικές προκειμένου να καταδεικνύονται οι περιφερειακές διαφορές στις ε, δημογραφικές εξελίξεις. Για αυτά τα θέματα μιλάμε πάντοτε. Επειδή η συχνότητα και η ποσότητα των στοιχείων που πρέπει να παρέχονται είναι ανοιχτή, ε, θα ήθελα αυτό εξ αρχής να γράφεται ξεκάθαρα. Για να μην πρέπει οι στατιστικές υπηρεσίες να επιβαρυνθούν με αδικαιολόγητα οικονομικά και διοικητικά εμπόδια. Ε, παράλληλα, θεωρώ σημαντικό κατά την ε, προετοιμασία των στοιχείων ε, να υπάρχει προστασία των προσωπικών δεδομένων. Γενικά δεν βλέπω μεγάλα προβλήματα και χαίρομαι που θα συζητήσουμε τις παρατηρήσεις σας και που θα συνεργαστούμε με τους σκιώδεις εισηγητές. Ευχαριστούμε πολύ. Ερίκα Μάνερ. Ευχαριστώ τον εισηγητή για την εξαιρετική του έκθεση. Η ομάδα μας μπορεί σε γενικές γραμμές να τον υποστηρίξω. Το πιο σημαντικό, το πιο σημαντικό θέμα είναι πώς στο μέλλον θα έχουμε τις λεπτομεριακές δημογραφικές στατιστικές και θα θέλαμε να γίνουν αυτές οι στατιστικές να είναι αξιόπιστες για την επιλεξιμότητα κάποιων ε, ε, σχεδίων, κάποια κονδύλια. Μας είπε η Κομισιόν ότι δεν είναι ακόμη πλήρως έτοιμες, αλλά θα πρέπει να μπορούμε να έχουμε αυτές τις στατιστικές, τις δημογραφικές για την κατανομή των κονδυλίων στη θέση μας. Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και τα προβλήματα κάθε περιοχής, να ληφθούν υπόψη ε, λεπτομεριακά. Γι' αυτό είμαστε υπέρ των προτάσεων αυτών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Προφανώς η Ευρώπη, όπως λένε οι στατιστικές, παρά το γνώσο ότι είναι λίγος υπάρχουν, έχει αυτό το πρόβλημα το δημογραφικό σε κάποιες περιοχές είναι πολύ σοβαρό. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ε, ως η συγγήτρια να συγχαρώ τη συγγήτρια και να πω τι γίνεται στη Γαλλικία. Στην, ε, στο κοινοβούλιο το τοπικό υπάρχει, δεδομένου ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα γύρανσης και έλλειψη στοιχείων και φεύγει ο κόσμος και έχουμε πολύ περισσότερα μεγάλα ε, άτομα τα οποία γυράσκουν παρά παιδιά που γεννιούνται, η ειδική επιτροπή που δημιουργήθηκε στο κοινοβουλίο μας. Εμείς ανήκουμε σε μια άλλη εποχή αν θέλετε. 20% όμως από τους ε, συναδέλφους μου που ήταν στο πανεπιστήμιο μαζί μου, της δικής μου γενιάς, ε, φύγανε από την περιοχή μας εδώ και 5, 10, 20 χρόνια και τώρα μένουν στο εξωτερικό και τώρα φεύγουν πολλοί νέοι. Πέρσι όταν δημοσιεύθηκαν ε, τα αποτελέσματα της πέμπτης έκθεσης ε, για τα θέματα αυτά τα κοινωνικά και την κατάσταση στις διάφορες περιοχές, στην έκθεση της συνοχής αναφερόταν από την Κομισιό ότι κάποια γεωγραφικά χαρακτηριστικά ή δημογραφικά θα μπορούσαν να οξύνουν ακόμη περισσότερο τα αναπτυξιακά προβλήματα. Στην Ευρω... περίπτωση της Ευρώπης, ακόμη και η έλλειψη εναρμόνισης κάνει απαραίτητο να έχουμε αυτό τον δείκτη δημογραφικής ε, ε, του ευάλωτου χαρακτήρα των ε, δημογραφικών. Γι' αυτό θα ήθελα να υποστηρίξω αυτό το οποίο είπε η συγγήτρια και να πω ότι τα μεγάλα και μόνιμα ε, μειονεκτήματα τα δημογραφικά θα πρέπει επίσης στην επόμενη προγραμματισμό να συμπεριληφθούν ως δείκτες. Γι' αυτό με μεγάλη ευχαρίστηση θα συνεργαστούμε με την εισηγήτρια. Ευχαριστώ. Ο κύριος Βανίστεροι. Και άλλη μια φορά δεν είναι εδώ η κυρία μου και να είναι, οπότε θα μιλήσω εγώ. Το 2012 είναι το ευρωπαϊκό έτος για την ενεργό γύρανση, την υγιή γύρανση. Το ότι γνωρίζουμε περισσότερες στατικές και κάνουμε λιγότερα βέβαια είναι πρόβλημα. Ίσως λοιπόν αυτό είναι ένα εργαλείο που θα μπορούσαμε και που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε. Είμαι θετικός λοιπόν ως προς τα όσα είπε η συγγήτρια. Περιμέναμε ότι θα είναι πολύ στοχευμένη η προσέγγιση. Απ' την άλλη, είναι περίεργο που αυτή τη στιγμή που έχουμε τη Eurostat και τόσο πολλά δεδομένα και νούμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και χρόνια, Πρέπει να έχουμε αυτό το δίκτυο δημογραφικής ευπάθειας. Προβλέψεις σε μια περιοχή όπου λέμε σε τι φάση βρίσκεστε ως προς τη γύρανση, πώς είναι οι νέοι. Ε, με αυτόν τον τρόπο γνωρίζουμε περισσότερα για την κατάσταση και τη θέση των ανθρώπων. Έτσι μπορούμε να αναπτύξουμε με περισσότερα κριτήρια αυτό το βασικό μοντέλο. Τέλος πάντων είναι σημαντικό ε, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο πρωταθλητής στη γύρανση. Έχουμε 20% του πληθυσμού που ε, μετά το που γυράσκει όντως κάτι συμβαίνει, τα πράγματα αλλάζουν ε, ως προς το χειρότερο συνέχεια. Ήμουνα σε μια συνεδρίαση της Επιτροπής Περιφερειών για τις κοινωνικές περιοχές και τι γίνεται με τις περιοχές όταν χάνουν τον πληθυσμό τους. Πραγματικά, πρέπει να υπάρξει αλλαγή στην προσέγγιση. Πρέπει να ενεργοποιήσουμε τις παλαιότερες γενιές και τις νεότερες γενιές. Είναι σημαντικό λοιπόν να μιλάμε για αυτά τα θέματα. Το ότι γνωρίζουμε περισσότερα δεν σημαίνει αυτόματα ότι κάνουμε και περισσότερα. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει στο πρόγραμμα περιεχόμενο που ε, να οδηγεί σε καινοτόμε ε, πολιτικές και σε εταιρικέ σχέσεις που θα μας βοηθήσει, μας βοηθήσουν με το στόχο του 2020. Ευχαριστώ. Σαμ Κέλλη. Ευχαριστώ. Συμφωνώ ότι προφανώς ε, ότι όσο πιο ακριβείς είναι στατιστικές είναι ακριβείς. Όσο πιο ακριβείς είναι οι στατιστικές, τόσο πιο εύκολο είναι κανείς να σχεδιάζει. Όμως, από την άλλη, το να συσσωρεύουμε στατιστικές ε, δεν έχει και πολύ αξία. Ε, τώρα, είτε είναι για την ε, ε, πολιτική συνοχή, για τη διακυβέρνηση, για την εκπαιδευτική, τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό, είτε τα γυμναστήρια, ας πούμε, όσο πιο ε, καλή είναι η συλλογή των στοιχείων, τόσο πιο εύκολη γίνεται η εφαρμογή σχεδίων που θα αντικατοπτρίζουν αυτά που θα συμβούν στο μέλλον σε επίπεδο δημογραφικό. Το δεύτερο σημείο που ήθελα να θίξω είναι αυτό που ανέφερε τελευταία ο εισηγητής, που έχει να κάνει με την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Φυσικά συμφωνώ με αυτό. Το συζητήσαμε σε πολλές συνεδρίες και χθε και σε άλλες που θα έρθουν. Η σημασία και η επικαιρότητα αυτού του θέματος είναι μεγάλη. Για τη συλλογή των στατιστικών τώρα, τι προσωπικά δεδομένα πρέπει να προστατευθούν. Ίσως θα πρέπει να σας εξηγήσω. Πρέπει να διασφαλίσουμε τα στοιχεία που έχουν να κάνουν να σας εξηγήσω ότι δεν μπορώ να καταλάβω. Μπορείτε να μας εξηγήσετε λίγο παραπάνω. Ναι, ευχαριστούμε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η Πρόεδρος θα καταλάβει ότι το θέμα της δημογραφίας ε, δεν με αφήνει διάφορο γιατί έχω πολύ καιρό έχω εργαστεί με τον Πρόεδρο Βερζές ε, που με έκανε ευαίσθητο ως προς την σημασία αυτού του θέματος. Συμφωνώ με τους άλλους ομιλητές. Είναι πολύ σημαντικό να μπορεί κανείς να έχει στη διάθεσή του πολύ συγκεκριμένα και ακριβή ε, δημογραφικά στοιχεία, ειδικότερα εφόσον υπάρχει αυτή η διαφορά μεταξύ των περιφερειών σε επίπεδο δημογραφικό. Από την άλλη υπάρχει μείωση του πληθυσμού στην Ευρώπη, ε, στις ε, ιδιαιτέρως απομακρυσμένες περιοχές για παράδειγμα. Θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας αυτή τη δημογραφική μετάφραση και αυτές τις δημογραφικές αλλαγές γιατί μπορεί ε, στο μέλλον να πρέπει να δεχθούμε χιλιάδες νέους κατοίκους, να βρισκόμαστε δηλαδή σε μια δύσκολη ε, θέση, σε μια αντίθετη τάση από αυτή που υπάρχει σήμερα στην Ευρώπη. Αυτά πρέπει να τα γνωρίζουμε με βάση τις ε, στατιστικές, γιατί μέχρι το 2050 λέμε ότι ο παγκόσμιος πληθυσμός θα είναι 9 με 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να έχει ένα πληθυσμό που μειώνεται και θα φτάσει στα 500 εκατομμύρια με επιπτώσεις σε όλους τους τομείς και φυσικά στην οικονομική ανάπτυξη. Έχω εδώ το νούμερο της Κομισιόν που λένε ότι τα συνδυασμένα, οι συνδυασμένες επιπτώσεις της δημογραφίας θα οδηγήσουν ε, στο να έχουμε μεταξύ του 2021 και 2031 2,1% μεγάλο πρόβλημα λοιπόν. Άλλο πρόβλημα είναι η επιβάρυνση στους ε, εργαζόμενους οι οποίοι ε, οι οποίοι αυτή τη στιγμή έχουν ε, πολύ μεγάλο δυσανάλογο αριθμό ηλικιωμένων να υποστηρίξουν. Αυτά πρέπει να ληφθούν υπόψη για τη λήψη πολιτικών αποφάσεων. Ευχαριστούμε πολύ. Ο Γιάνν Όλμπριχτ. Ναι. Νομίζω ότι συζητούμε τα νομικά προβλήματα και φυσικά υπάρχει μια συνεχής ε, συζήτηση μεταξύ των δημογραφών, των υπεύθυνων για τη δημογραφία που αναρωτιούνται τι είναι τα στοιχεία που πρέπει να συλλέξουν. Υπάρχει και το θέμα της ε, συνοπτικής παρουσίασης των στοιχείων. Ποια είναι τα στοιχεία που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε, πώς θα τα συγκλέξουμε, σε τι επίπεδο, πώς θα τα συγκεντρώσουμε, πώς θα διασφαλίσουμε την ε, συνεργασία μεταξύ των διαφόρων επιπέδων με αυτή την συγκέντρωση των στοιχείων. Τι θα γίνει, πρέπει να αλλάξουμε κάτι. Αναφέρω αυτά που υπόθηκαν χθε ε, στην συνάντηση του ΩΣΑ, όπου αναφέρθηκε ότι πρέπει ε, να υπάρξει αλλαγή του τρόπου συλλογής στοιχείων και στην Ευρώπη. Για μένα είναι σημαντικό, γιατί στη δική μου έκθεση θα προτείνω να ε, διευρυνθεί το πεδίο παρέμβασης για περιοχές στις οποίες υπάρχουν προβλήματα λόγω δημογραφικών εξελίξεων. Γι' αυτά θα χρειαστούμε πολύ ξεκάθαρα στοιχεία. Γι' αυτό νομίζω ότι αυτή η έκθεση ε, σχετίζεται άμεσα με το ΕΣΠΑ και αν δεν έχουμε ξεκάθαρα στοιχεία, το ΕΚΠΑ, συγγνώμη, και αν δεν έχουμε ξεκάθαρα στοιχεία δεν θα μπορέσουμε να έχουμε... Ξέρω αν υπάρχει κάποιος από την Κομισιό που θέλει να λάβει το λόγο. Η κυρία Κλεμονσό έχει το λόγο. Thank you Από την Επιτροπή και την Eurostat ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον εισηγητή και τον ε, για την ε, έκθεση και την υποστήριξη. Η Eurostat και η Επιτροπή συλλέγουν εδώ και πολλά χρόνια δημογραφικά δεδομένα και τα συλλέγουν σε εθνικό τοπικό επίπεδο ακόμη έχουμε προβλήματα συγκριτικής ανάλυσης και δεν είναι πάντα σαφή τα στοιχεία που έχουμε από όλους. Θα πρέπει λοιπόν την συγκρισιμότητα αυτών των δεδομένων να τη βελτιώσουμε. Γι' αυτό το ρόγο, με τον κανονισμό αυτό, θέλουμε, όπως είπατε και στην έκθεσή σας, να ορίσουμε τον τόπο διαμονής, τον κύριο τόπο διαμονής των πολιτών για να ξέρουμε πού ανήκουν. Στη Ρουμανία, Φερρυπίν, υπάρχουν άτομα τα οποία στις απογραφές καταγράφονται ενώ ζουν 10 χρόνια στο εξωτερικό και δεν θα πρέπει σύμφωνα με τον ορισμό της συνήθους τόπου διαμονής να καταγράφονται. Τέτοιου είδους προβλήματα λοιπόν θέλουμε να ξεπεράσουμε και με αυτόν τον κανονισμό θέλουμε να βελτιώσουμε τη συγκρισιμότητα των δεδομένων. Επαναλαμβάνω και να έχουμε λεπτομεριακά στοιχεία σε περιφερειακό, τοπικό, εθνικό και γενοτικό στοιχείο και να έχουμε και άλλους δείκτες. Καλύτερα και περισσότερα δεδομένα ώστε να μπορούμε να έχουμε πιο αξιόπιστους δείκτες. Αυτός είναι ο στόχος μας. Θα ήθελα τώρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων να πω ότι με αυτό τον κανονισμό μιλούμε για ενοποιημένα στοιχεία τα οποία αποστέλλονται σε μορφή πίνακα. Δεν πιστεύω λοιπόν ότι υπάρχει κίνδυνος σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα, γιατί είναι ενοποιημένα. και αφορούν ε, ε, τα άτομα ανα κατηγορίες, ανα φύλλο, ανα έτος, γέννης κτλ, κτλ. Δεν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος. Λοιπόν, ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Η Ευχαριστώ λίγο σύντομα γιατί μετά από την ανταλλαγή απόψεων έχω κάποια σχόλια να πω ότι πρόκειται για έναν τεχνικό κανονισμό και το πώς θα χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα είναι κάτι που θα πρέπει να το συζητήσουμε στην πρωτοβουλία, όμως που είχαμε τα τελευταία χρόνια με μια έκθεση. Εκεί αναφέρεται ότι ε, πρέπει να έχουμε συλλογή στοιχείων ακριβώς για τα πράγματα για τα οποία να, μιλήσατε. Για να μπορούμε όχι μόνο να συγκρίνουμε μεταξύ τους περιφέρειες, αλλά να μπορούμε στην ίδια την περιφέρεια να πάμε και να δούμε πώς διαμορφώνονται οι διαμογραφικές εξελίξεις και έτσι να μπορούμε να έχουμε συγκεκριμένα στοιχεία. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να τα παρακολουθούμε όλα αυτά στο Δινεκές, γιατί εμείς εδώ στο Κοινοβούλιο έχουμε ως καθήκον να βρίσκουμε τις αντίστοιχες λύσεις και χρειαζόμαστε τα κατάλληλα δεδομένα για να μπορούμε να βρίσκουμε όλες αυτές τις κατάλληλες λύσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Κλείνει η συζήτηση. Η προθεσμία για τις τροπολογίες είναι και αυτή σύντομη. 22 Ιουνίου στις 12 μετά μεσημβρίας εξαιτία του γεγονότος ότι η ψηφοφορία στην Επιτροπή είναι πριν από τη δική μας ε, το Σεπτέμβριο, οπότε πρέπει να ψηφίσουμε τον Ιούλιο. Τελειώνει η σημερινή συνεδρίαση. Πάμε στη συνάντηση των συντονιστών. Καλέσαμε τους πράσινους πριν από λίγα λεπτά, γιατί μόνο αυτοί μας λείπουν και δεν ξέρω αν είναι εδώ. καφέ, ναι. Καλό είναι ο καφές. Εντάξει, να έρθουν οι συνάδελφοι και ξεκινάμε τη συνάντηση των συντονιστών. Μπορεί κάποιος να δει ποιοι πίνουν καφέ. Thank you.